and I think it will work. Okay. Looking for a fairy godmother. The first time I uh, have such experience. Μας ακούτε. Εσείς μας ακούτε. Καμία καμπίνα δεν ακούει τίποτα από την αίθουσα. Περιμένω. comprendre. Περιμένουμε να λυθεί λοιπόν αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Λυπούμαστε πάρα πολύ, αλλά καμία καμπίνα δεν ακούει τίποτα από την αίθουσα, από όσα διαμείβονται. Για να δούμε Λοιπόν, μου λένε ότι είναι εντάξει. Είναι εντάξει τώρα, μάλιστα. Είναι εντάξει, τώρα ακούμε. Επιτέλους, ναι, ναι. Ε, και στα Ιταλικά, διερμηνία και απ' όλα. Είμαστε εντάξει. Ιταλικά έχουμε. Ελληνικά και πάλι τελευταία δοκιμή, τώρα λειτουργούν μάλλον όλες οι γλώσσες. Εντάξει, τώρα ακούμε από την αίθουσα, έχουμε ήχο. Ευχαριστώ πολύ. Κιθ. Και τώρα μπορείς να συνεχίσεις από εκεί που σταμάτησες ή να ξαναρχίσεις όπως θέλεις. Make you sit through it all again. Um, I was wanting to mention why I was doing this report. Να μην τα ξαναπώ από την αρχή, να σας πω γιατί κάνω αυτή την έκθεση. Εξηγούσα ότι η έκθεση πραγματεύεται με τα μέτρα έτσι ώστε ο κλάδος των πλωτών επιβατικών μεταφορών να είναι ε, πιο ανταγωνιστικός, πιο καθαρός, πιο πράσινος και πιο φιλικός και προς τα κοινωνικά και προς το περιβάλλον και να εξασφαλίζονται και τα δικαιώματα των ε, επιβατών ε, στις θαλάσσιες μεταφορές και στις εσωτερικές πλωτές οδούς. Άρα να βελτιωθεί και η ποιότητα των υπηρεσιών και η προσβασιμότητα του κλάδου. Σας ευχαριστώ για τις τροπολογίες σας αγαπητοί Σκιώδης. Ε, συμβιβαστική αν αναφέρθηκα ήδη σε αυτή και όπως είπατε τόσο ωραία και συμφωνήσατε, θα πάω αμέσω στη συμβαστική υπαριθμό 2 που εξασφαλίζει το γεγονός ότι η παράγραφος 5 να τονίζει επίσης το πλεονέκτημα της αποσυμφόρησης των οδικών μεταφορών και των χερσαίων γενικά, ε, έτσι ώστε να έχουμε ε, πλωτές ε, μεταφορές και σε συνδυασμό με τις ε, αστικές και περιστικές συγκοινωνίες. Οι επενδύσεις θα πρέπει να αφορούν την ποιότητα των υποδομών και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ένα κατάλογο καλών πρακτικών στον τομέα αυτό. Επιπλέον, υπάρχει ε, πολύ ε, μεγάλη σημασία για την κατάρτιση και τις μεθόδους κατάρτισης σε ε, συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοίας ΑΕΜΟ και τον ILO έτσι ώστε να υπάρχει και ε, μια σύνδεση ανάμεσα στην ποιότητα, την ασφάλεια και το καταρτισμένο προσωπικό έτσι ώστε ε, να ε, είναι ασφαλής ο τομέας αυτός. Αυτό το λέμε στην Συμβαστική 3. Θα πρέπει να αναπτυχθεί ο βιώσιμος και αηφόρος τουρισμός και αντίστοιχα η τροπολογία Συμβαστική 4 κάνει λόγο για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες και περιφερειακές περιοχές της Ένωσης και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ε, τη χρήση των ε, κοινωτικών κονδυλίων. Και συμβαστική 5, ε, τηολογική σκέψη Β, τονίζει τη σημασία των πλωτών μεταφορών επιβατών στη διασύνδεση των διαφόρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που συνεισφέρει προς την ενίσχυση της συνοχής και ανταποκρίνεται και από τι αναφόρο τιμής στις τεχνολογικές εξελίξεις και στο σχεδιασμό των σκαφών. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένω να ακούσω τους σκιώδεις και να εγκριθεί η έκθεση αύριο το πρωί στην Επιτροπή μας. Ελπίζω να ε, οθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να δράσουν γρήγορα και να έρθουμε ένα βήμα πιο κοντά στο να γίνει πραγματικότητα το τεράστιο δυναμικό των πλωτών μεταφορών για να μειωθεί η συμφόρηση, επαναλαμβάνω, ε, των ε, δρόμων μας και να μειωθεί και η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τέιλορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να προσθέσω πολλά σε όσα είπε ο εισηγητής. Πιστεύω ότι η έκθεση είναι ιδιαίτερα ισόρροπη και πολύ καλά διορθωμένη και διεξοδική. Με πέντε συμβαστικές τροπολογίες που μπορούμε να συμμεριστούμε και εκφράζουν συνολικά την πρόθεση της επιθυμίας των περισσότερων σκιωδών στο θέμα αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε καλό αποτέλεσμα. Στηρίζουμε λοιπόν το έργο του Σκιώδους, του εισηγητή, συγγνώμη, και Απλώ δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να έχουμε και έναν οργανισμό για την εσωτερική ναυσοπλοεία στην Ευρώπη. Εκεί υπάρχουν πολλέ τροπολογίε, μία από τι οποίε και τη δική μου ομάδα. Απλώ να ε, ρωτήσω τι θα γίνει με την τροπολογία 85. Εκεί έχω μια απορία. Ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο εσωτερικό των κρατών μελών να προωθήσει την υιοθέτηση μέτρων φορολόγησης για τους φορείς προκειμένου να βελτιώσουν το σύστημα ασφάλειας στα σκάφη της εσωτερικής ναυσιπλοείας. Είναι η ασφάλεια μια προτεραιότητα βέβαια, αλλά αυτό θα μπορούσαμε να το πετύχουμε με πολιτικές που να προσφέρουν κίνητρα, όπως αυτές που σκοπό έχουν να στηρίξουν γενικότερα τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ο κύριος Κύρκος παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Τέιλορ και τους υπόλοιπους ε, και τους σκιώδεις εισηγητές. Πραγματικά καταλήξαμε σε πέντε τροπολογίες οι οποίες ε, ενδυναμώνουν την ε, πραγματικά ενδιαφέρουσα το ενδιαφέρον Initiative Report. Ε, αν είχα να κρατήσω δύο-τρία πράγματα από τις συζητήσεις που κάναμε ήταν το ιδιαίτερο βάρος που θέλουμε να δώσουμε στην υποβοήθηση των περιφερειών και των παραμεθόριων περιοχών, όπως είναι τα ελληνικά νησιά, τα Κανάρια, οι Αζόρες και πώς οι θαλάσσιες μεταφορές, οι πλωτές μεταφορές επιβατών πρέπει να μην υποβοηθούνται μόνο κατά τη διάρκεια των τουριστικών περιόδων αλλά και γενικότερα γιατί είναι ε, μια, ένας πόρος ζωής για αυτές τις περιοχές για το θέμα της ε, ασφάλειας τονίσαμε πόσο σημαντικό είναι, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πάρουμε μέτρα ώστε να μην οποιαδήποτε κίνηση στον τομέα της ασφάλειας που είναι υποχρεωτική να μην εμποδίσει την ε, φυσιολογική και σωστή και γρήγορη ροή ε, επιβατών και εμπορευμάτων. Επίσης ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι διευρύναμε το πεδίο εφαρμογή της έκθεσης, αλλάζοντας και τον τίτλο από εκεί που ξεκινούσαμε μόνο για τα πορθμία, τώρα βάλαμε μέσα και, τις, και την κρουαζιέρα που σε θέματα όπως είναι ε, το περιβάλλον, ας πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να, βάλουμε, να πάρουμε υπόψη και τα μεγάλα σκάφη της κουραζιέρας. Επίσης και οι δυνατότητες δανειοδότησης και εγγυήσεων για τα έργα των πλωτών μεταφορών που έρχονται και από το ε, EFSI μαζί με όλα τα άλλα. Εν ολίγης πιστεύω πως έχουμε μια πολύ προσεγμένη και ισορροπημένη έκθεση και προσλέπω και εγώ στην ψήφισή της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για τον ε, Κίθ. Πραγματικά ήταν πολύ ευχαριστή η δουλειά που κάναμε σε μια πολύ θετική ε, έκθεση, η οποία ε, ήδη από την αρχή συγκέντρωνε σε ευρεία συνένεση. Γνωρίζουμε βέβαια όλοι πόσο σημαντικές είναι θαλάσσιες μεταφορές και υπάρχουν πολλές επιτυχίες με τις οποίες συμφωνούμε όλοι μας σε αυτή την εκθέση. Δηλαδή θα πρέπει να έχει χαρακτήρα φιλικό προς το περιβάλλον, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στη διασύνδεση ειδικότερα των απομακρυσμένων περιοχών. Οπότε όλοι συμφωνούμε με αυτέ τι συμβαστικέ τροπολογίε. Οπότε δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η Άλντε έχει βγει από τη συμβαστική τροπολογία 5. Εμεί είπαμε ότι συμφωνούμε με όλε αυτέ τι συμβαστικέ τροπολογίε. Ε, θα υπερψηφίσουμε λοιπόν και την 5. Ε, ε, αλλά δεν περιλαμβανόμαστε τουλάχιστον στο voting list αυτή τη στιγμή. Αλλά σα λέω από τώρα η Άλτε θα υπερψηφίσει τη συμβαστική 5. Επίση, ε, εμείς θεωρούμε πως δεν χρειαζόμαστε μία νέα υπηρεσία, μία νέα αρχή, γιατί ήδη υπάρχει σε διεθνές επίπεδο η IMO, ο διεθνέ Αυτιλιακός Οργανισμός, και από εκεί και μετά υπάρχει η ΣΕΣΝΗ, Επιτροπή δηλαδή των ε, οι διάφορε επιτροπέ ε, ποταμών. Οπότε, καλό είναι βέβαια και θετικό ακούγεται να λέμε ότι θα εστιάσουμε σε ένα συγκεκριμένο τομέα, επειδή ακριβώ οι πλωτέ μεταφορέ συχνά ε, δεν βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντο. Συχνά λοιπόν ε, είναι θετικό το να λέμε ότι θέλουμε κάτι καινούριο, αλλά υπάρχουν ήδη εδώ μια σειρά από φορεί, οπότε δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερου. Απλώ θα πρέπει να εστιάσουμε καλύτερα τι προσπάθειε, να έχουμε μια καλύτερη υποπτία και μια καλύτερη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των υφισταμένων αυτών οργανισμών. Πάντω, ε, κατά τα λοιπά, ε, συμφωνώ με όλες τις ε, πτυχές, συμφωνώ με αυτή την έκθεση και πραγματικά πολύ καλή δουλειά που κάναμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, ευχαριστούμε και για όλα αυτά τα θετικά σχόλια, είναι θετικό αυτό το γνώμη και σημειώνουμε πράγματι ότι υποστηρίζει άλλη, και τη συμβαστική τροπολογία 5. Αυτό για αύριο για την ψηφοφορία. Τάνια Κουζάλη πέντε τώρα, επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για τη δουλειά του. Έχει την καλοσύνη ε, να επιδείξει πνεύμα συνεργασίας και επικοδομητικό κατά τη διάρκεια της εκπόνησης έκθεσης. Και πιστεύουμε ότι αύριο μετά την ψηφοφορία η έκθεση θα είναι ισορροπημένη και καλή και στην ίδια γραμμή που έχουμε εργαστεί εδώ και καιρό στην Επιτροπή μας για να προωθήσουμε τις μεταφορές πιο αποτελεσματικές και πιο βιώσιμες που θέλουμε. Η έκθεση αυτή είναι ένα πρώτο βήμα. Ξεχάσαμε όμως κάποιες αποχρώσεις που θεωρούμε σημαντικές και ακόμα δεν έχουν επιληθεί που ενδεχομένως θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι τη διαφορά εμείς ε, όταν θέλουμε να κάνουμε μια καλή πολιτική μεταφορών. Παράδειγμα, διαφοροποίηση ανάμεσα στους διάφορους τύπους σκαφών και αποστολή τους. Μιλάμε για επιβατικές μεταφορές, θαλάσσιες και ποτάμιες, αλλά δεν είναι το ίδιο το πορθμίο με το κουρασγερόπλιο, πούμε, ούτε είναι η ίδια ε, ζημιά που κάνουν στο περιβάλλον. Ε, άλλο είναι ένα δρομολόγιο, μια ακτοπλοεία, ας πούμε, ή ε, μικρά σκάφη που με ένα καλό σχεδιασμό μπορεί να είναι βιώσιμη ε, μορφή ε, έτσι, κανονικής κυκλοφορίας και άλλο είναι κάτι θηρία κρουαζιερόπλια που έχουν αναψυχή ως στόχο και περιοδικό χαρακτήρα. Μιλάμε για τη βιώσιμη ε, ανάπτυξη και του αεροπλάνου και του αυτοκινητόδρομου σε συνδυασμό με τις πλωτές μεταφορές, αλλά δεν μιλάμε για τον οικονομικό αντίκτυπο, τον κοινωνικό, ούτε τον περιβαλλοντικό. Ούτε τα πιο απλά δεν λέμε, δηλαδή πώς μπορεί ε, να δοθεί νέος δυναμισμός αποκεντρωμένος στην περιφέρεια με τα ποτάμια, αυτό συνεισφέρει στην εδαφική και στην κοινωνική συνοχή, μακροπρόθεσμα και θα έχει και αντίστοιχη ε, απόδοση περιβαλλοντική. Δεν μιλώ μόνο για καυσαέρια εδώ και αέρια του θερμοκηπίου, αλλά και για ρήπανση των υδάτων και τα στερεά απόβλητα. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είναι καλή, είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά να έχουμε επίγνωση ότι χρειάζονται και άλλα ακόμα βήματα πολλά να γίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλο ομιλητή. Η DigiMove, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Κριστίνα Μπέρκ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής σας για αυτή την πρωτοβουλία. Την καλωσορίζουμε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι θεωρούμε ότι δεν είναι απλώς ισορροπία, αλλά είναι και επίκαιρη. Θα γνωρίζετε ίσως ότι η Επίτροπος Μπούλτς υπεύθυνη για τι μεταφορές, αποφάσισε το 2017 να γίνει το ευρωπαϊκό έτος για τις εσωτερικέ και τι πλωτέ, μάλλον μεταφορές. νομίζω εννοείται 17, όχι 70. Ναι, χαχα. Ε, ναι, μιλάμε λοιπόν για τις πλωτές μεταφορές και νομίζω ότι με την έκθεση αυτή το Κοινοβούλιο προλαμβάνει τις εξελίξεις κάτι πολύ θετικό. Ε, για μερικά επιμέρους ζητήματα σε σχέση με την όλη συζήτηση που είχαμε και συγκεκριμένα τις συμβιβαστικέ τροπολογίες, κατά πρώτον νομίζουμε ότι ίσως να έχει κάποιο νόημα να κάνουμε διάκριση μεταξύ μεταφορών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων όπως οι κρουαζιέρες, είτε είναι στη θάλασσα είτε σε ποτάμια που σίγουρα δεν έχουν τον ίδιο ρόλο στην διασύνδεση διάφορων περιοχών μεταξύ τους, στις εξόχως απόκεντρες, ε, στην δημιουργία συνοχής, καθώς και τους όλους προβληματισμούς για το πώς να διευκολύνουμε αυτό το είδος τις μεταφορές λόγω χάρη με υποχρεώσει όπω για τι δημόσιε υπηρεσίε. Εκεί θα είναι διαφορετικέ υποχρεώσει όταν μιλάμε για κρουαζιέρε, τουριστικέ κρουαζιέρε, μια ανθούσα ε, επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν χρειάζεται αυτή η καθεαυτή στήριξη. Σε ό,τι αφορά την προστασία των εξωτερικών συνόρων και με όλα τα θέματα που μας απασχολούν σε σχέση με την ασφάλεια, η Επιτροπή εκτιμά το ρόλο της Επιτροπής σας και προσφάτως στην ενίσχυση του Οργανισμού για την ε, ασφάλεια, τη θαλάσσια ασφάλεια και σε συνεργασία με τη Frontex και την, ε, τον οργανισμό της Αλίας των αλληλευτικών δραστηριοτήτων, ώστε να διασφαλιστούν τα εξωτερικά σύνορα, να, ε, να αντιληφθούν οι σχετικές πληροφορίες και να έχουμε μια συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει στις θάλασσές μας. Κάτι πολύ σημαντικό, ένα βήμα που οπωσδήποτε ε, έπρεπε να αντικατοπτρίζεται και αυτό στην έκθεσή σα. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά δεδομένα, στατιστικά δεδομένα που είναι πολύ σημαντικά για την ανάλυση του τι συμβαίνει ως προς αυτήν την μορφή των επιβατικών μεταφορών, στηρίζουμε την έκκληση να συγκεντρώνονται περισσότερα στατιστικά στοιχεία, όμως να θυμίσουμε ότι η Eurostat δραστηριοποιείται στη συλλογή τέτοιου είδους δεδομένων μόνον εφόσον το ζητά, το απαιτεί η νομοθεσία. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προπαρασκευαστική φάση θα έπρεπε να αποτεμήσει το διοικητικό άχθος προς τους ε, ενδιαφερομένους φορείς για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών. Ένα καμπόδε ζήτημα από μόνο του για να ζητηθεί κάτι τέτοιο από την Eurostat. Ε, κλασικά, ε, παραδοσιακά, μάλλον ο στόχος είναι η μείωση των δεδομένων που συγκεντρώνονται και όχι το αντίστροφο. Πάντω, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επειδή μιλάμε για ένα έτο για τι θαλάσσιε μεταφορέ, θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε τι επιχειρήσει που ασχολούνται με κρουαζιέρε και να δούμε κατά πόσον μπορούμε να έχουμε μαζί του μαζί τους μια συνεννόηση για στατιστικά στοιχεία και για πληροφορίε για το τι συμβαίνει στου επιμέρου λιμένες. Αυτό έστω προσωρινά, ώστε να υπάρξει νομική βάση για να συγκεντρώνει περισσότερα δεδομένα η Eurostat. Να δούμε μήπως οι εταιρείε μπορούν να μας δίνουν περισσότερες σχετικές πληροφορίες. Επίσης υπάρχει αυτός ο πολύ σημαντικός τομέας όπου συλλέγουμε δεδομένα για ατυχήματα. Εκεί βασίζονται όλες οι δραστηριότητέ μας σε σχέση με την ασφάλεια. Εδώ είναι σχετικά δυσάρεστο που ο Οργανισμός για τι Θαλάσσιες Μεταφορές, ε, βάσει της οδηγίας για τα θαλάσσια ατυχήματα και τις ερευνές τους, δεν συγκεντρώνει δεδομένα. Υπάρχει μια ετήσια έκθεση, η οποία είναι πολύ ε, σκόπιμη, πολύ εύστοχη μάλλον, ε, τη συνιστώ προς ανάγνωση, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για την εσωτερική ναυσιπλοεία ακόμα. Ως προς το σύνολο του συνδυασμού των διαδρομών εσωτερικής ναυσιπλοείας, με άλλους τρόπους μεταφοράς. Συμμεριζόμαστε τις απόψεις σας ότι αυτό μπορεί να είναι ε, απλώς και μόνο εποφελές. Πολλά γίνονται βάσει τις οδηγίες ITS για την, ε, συγκεκριμένη, για την ενιαία έκδοση εισιτηρίων, γιατί σε αυτό το πλαίσιο θα μπορεί κανείς να αγοράσει ένα εισιτήριο και μετά με αυτό το εισιτήριο να συνεχίσει λόγου χάρη με ένα επιβατικό ε, σκάφος. Υπάρχουν πολλά στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι είναι καλό να γίνουν τέτοιοι συνδυασμοί. Ε, μέχρι το 2019 το ίδιο και τα χρονοδιαγράμματα των διαφορετικών ε, ταξιδιών και διαδρομών, καθώς και οι σχετικές και σκόπιμες πληροφορίες για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Βεβαίως, όλοι συμφωνούμε ως προς τη σημασία του ΑΕΜΟ και του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας δηλαδή το ρόλο του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοείας και του ε, Οργανισμού Εργασίας, ε, ο Οργανισμό Ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ήδη εντατική δουλειά για το πώ ε, εφαρμόζονται όλε αυτέ οι διατάξει. Δεν έχουμε βέβαια ειδικό οργανισμό για του δρόμου τη εσωτερική ναυσιπλοεία. Αν δημιουργεί το τέτοιο οργανισμό, θα υπήρχε πρώτα απ' όλα θέμα για τον προπολογισμό. Ίσως και το Κοινοβούλιο να θέλει να ξανασκεφτεί αυτές τις πτυχές και ως προς τις συζητήσεις που γίνονται για το ερχόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις προοπτικές του. Με αυτά και με αυτά θα ήθελα να ολοκληρώσω και να επιστήσω την προσοχή σας σε μια πρόσφατη έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 30 Σεπτεμβρίου τρέχοντος. Εκεί ε, παρουσιάζεται η αποτίμηση της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αυσιπλοεία 2009-2019 με όλες τις πληροφορίες για την εσωτερική ναυσιπλοεία και για τις πέντε περιοχές προτεραιότητας, βιωσιμότητα, ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα, και έχει αποσταλεί και στη γραμματεία σας προς ενημέρωση. Ελπίζω να σας ε, την μοιράσουν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για το γεγονό ότι διανεμήθηκε, πράγματι το γνωρίζουμε και δίνω και πάλι για να κλείσουμε αυτό το θέμα τον ε, λόγο στον Κίχτέλο. Ε, σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Ε, Κούτερα και εσύ κάποιος άλλος συνάδελφος, δεν θυμάμαι τον. Επίσης, αφού άκουσαν ε, και τα όσα είπαν οι σκιώδεις, ότι πράγματι ε, χρειαζόταν παραπάνω σκέψη ό,τι αφορά αυτόν τον ε, οργανισμό. Και είναι ενδιαφέρον το ότι ακούσαμε μόλι τώρα από την Επιτροπή να μα λέει ότι πράγματι η δημιουργία ενό τέτοιου οργανισμού εξαρτάται από τον προπολογισμό, από τα κονδύλια. Ε, Ενδεχομένω, δηλαδή μπορούμε προ το παρόν να επιτύχουμε τον κατάλληλο έλεγχο τη κατάσταση βασιζόμενοι στι εφιστάμενες ε, αρχέ υπηρεσίε. Επίση, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα διαφορετικά είδη, στου διαφορετικού τύπου ε, πλοίων. Και ότι αυτές, αυτοί οι διαφορετικοί τύποι δημιουργούν διαφορετικές ευκαιρίε, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα τακτικά πορθμία. Για παράδειγμα εδώ αναφέρομαι σε κάποια παραδείγματα στη Δανία, αλλά και στο Άμστερνταμ, όπου έχουμε για παράδειγμα ηλεκτροκίνητα τέτοια απορθμία φέρει, τα οποία ε, ε, παράγουν πραγματικά πολύ περιορισμένη μόλις. Τέτοιου είδους λοιπόν τεχνολογίες αποτελούν μια ευκαιρία και γνωρίζω πως η Επιτροπή ε, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την ανάπτυξη τέτοιου είδους πρωτοβουλειών χαμηλών εκπομπών άνθρακα. γιατί βέβαια με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στο επίπεδο της κλιματικής αλλαγής και βέβαια ε, ταυτόχρονα βοηθούν την αποσυμφόρηση των οδικών μεταφορών. Χαίρομαι λοιπόν ε, για το γεγονός ότι το 2017 ε, μπορεί να είναι αυτό το έτος για την σε μεταφορές, γιατί πραγματικά θα πρέπει όσο είμαστε ακόμα εδώ σε, την, ε, σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο εμείς ως πράσινοι να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Πρόεδρος, αύριο λοιπόν είναι η ψηφοφορία για αυτό το ζήτημα, οπότε περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά δηλαδή το ρόλο του αλλιευτικού τουρισμού ε, ε, σε ό,τι αφορά την προώθηση του τομέα της αλληλείας έχουμε να δώσουμε κατευθείαν το λόγο στον κύριο Ινωή που είναι ο εισηγητής για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης ε, προσπαθώ να απαντήσω ένα βασικά ερώτημα. Πώς ε, μπορεί ο κλάδος της αλληλείας να επωφεληθεί από τον ελευτικό τουρισμό για να διαφοροποιηθεί ε, περισσότερο. Πώς μπορούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε ε, θέσεις εργασίας με ένα βιώσιμο τρόπο, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους εργαζόμενους σε αυτό το τομέα να διατηρήσουν την ταυτότητά τους ε, και την παραδοσιακή τους απασχόληση. Υπάρχουν κάποια εξαιρετικά παραδείγματα σε ορισμένες χώρες, όπως την Ιταλία, στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία και ειδικότερα σε και παράκτη δραστηριότητε αλλά ε, υπάρχει η πρόθεση να ε, συμπεριληφθούν περισσότερο και οι εσωτερικές ε, οδυναύσεις Για παράδειγμα, οι λίμνες και οι ποταμοί. 74 συνολικά τροπολογίες υποβλήθηκαν και επειδή η πλειοψηφία τους περιλάμβανε νέες ιδέες, θεώρησα πως δεν χρειαζόταν συμβαστικέ τροπολογίε, αλλά τελικά για να ενοποιήσω καλύτερα το κείμενο αποφάσισα να προτείνω τέσσερι συνολικά συμβαστικέ τροπολογίε. Η πρώτη από αυτέ προσπαθεί να επιτύχει τον καλύτερο δυνατό τουρισμό του αλευτικού τουρισμού. Δηλαδή, ε, περιλαμβάνουμε τον ε, τουρισμό Πέσκα και ήτη, όπω ε, με ενημέρωσε σε κάθε περίπτωση ο Ιταλό συνάδελφο. Και εστίαση στις συνέργειες σε αυτό το κλάδο για ε, την ε, δημιουργία ε, προϊόντων υψηλής ποιότητας σεβόμενη την ε, κληρονομιά σε αυτού ε, του τομεί και την ε, διαφοροποίησή του. Η δεύτερη συμβαστική τροπολογία αναφέρεται στο γεγονό ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν πλατφόρμε marketing, προώθηση δηλαδή στην αγορά, οι οποίε θα ανταποκρίνονται στι συγκεκριμένε ανάγκε για αυτά τα προϊόντα. Η τρίτη συμβαστική τροπολογία αναφέρεται στο ζήτημα τη βιωσιμότητα και στην σημασία του να υπάρχουν επιχειρησιακά μοντέλα που είναι ακριβώ φιλικά προ το περιβάλλον. Και εδώ τονίζεται και ο ρόλο που καλούνται να παίξουν οι εμπειρογνώμονε σε ζητήματα προστασία του περιβάλλοντο. Στην τελευταία συμβαστική τροπολογία καλούμε την Επιτροπή να αξιοποιήσει με τον εντεδειγμένο τρόπο τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα ε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Θάλασσα και την Αλία, ειδικότερα για τη μετασκευή και για τον εξυγχρονισμό ε, των ε, σκαφών της επαγγελματική αλίας. Εκεί καλούμε και την Επιτροπή να παρέχει σε περιφερειακό επίπεδο τις κατέλεσε πληροφορίε στα κατάλληλα δεδομένα και σε τακτά χρονικά διαστήματα μα ενημερώνει ω προ το ποια project έχουν λάβει χρηματοδοτική υποστήριξη και σε ποιο βαθμό, πια κονδύλια δηλαδή. Ε, θεωρούμε πως ε, έχουμε κάνει λοιπόν μια πολύ καλή πρόοδο, φτάνοντας σε ένα πολύ καλά διατυπωμένο και ισορροπημένο κείμενο. Αν έχετε άλλες προτάσεις θέλω να τις ακούσω. Για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εργασία που κάναμε, γιατί όπως γνωρίζετε εγώ είμαι από την Ουγγαρία και η δική μου χώρα δεν έχει πολύ ε, θάλασσα αν θέλετε. Οπότε πραγματικά ήταν για μένα πολύ εντακτική αυτή η εργασία. Σίγουρα όμως ε, πραγματικά πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο όπως αναφέρουμε και στην εκθέση στους, ε, στις, λιμένες και στις, ε, στις, λίμνες συγγνώμη, και στους εποταμούς. Ναι, λέει ο πρόεδρος, αλλά έχουμε και το, έχετε το Δούνα, μην το ξεχνάτε αυτό. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Η συνάδελφός μου, η κυρία Σουίτσα, είναι καθοδόν ακόμα ε, για να φτάσει στις Βρυξέλλες δεν έχει εφηχθεί ακόμα και μου ζήτησε να πω δύο λόγια εξ ονόματός της και ε, προς τον ε, εισηγητή μας. Τώρα είπατε για το Δούναβι στην Ουγγαρία, αλλά υπάρχει και η λίμνη Μπαλατών που είναι πάρα πολύ ωραία για να κυκλοφορούν εκεί τουριστικά και αλευτικά σκάφη. Είναι ιδεώδης συνδυασμός. Είναι πάρα πολύ καλή αυτή έτσι κι αλλιώς η πρωτοβουλία κατά την άποψή μου και ε, ε, η, η Αλία ε, όλο ασχολείται με τα αλλιευτικά πεδία και με την απόδοση. Αν μπορεί να συνδυαστεί με τον τουρισμό η Αλία, είναι ένα καταπληκτικό μοντέλο. κατάλαβα ότι υπάρχουν τέσσερις συμβαστικές τροπολογίες. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συμφωνεί απολύτως και υπερψηφίζει και ελπίζω αύριο το πρωί να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή και να περάσει. Και πάλι ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή μας ε, για να στείλουμε και στην Επιτροπή Αλίας και τη δική μας άποψη και τους θορύβους και τους ψηφίρους από τις μεταφορές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Γεζίνε Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και τον αγαπητό συνάδελφο από την Ουγγαρία που μόλις μάθαμε ότι ψαρεύετε κιόλα εσύ, εσύ εκεί ε, από τη γνωμοδότησή σας. Ε, θέλω να σας πω ε, ότι προεξοφλούμε συμφωνία από τους φιλελευθέρους και για τις τέσσερις τροπολογίες. Είναι σημαντικό να έχουμε μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Αλίας, γιατί μπορεί να μην τους πέρασε από το μυαλό ότι η Αλία έχει να κάνει μεγάλη σχέση με τον τουρισμό. Και όσοι ζουν σε παραθαλάσσιες περιοχές και ψαροχώρια, εν πάση περιπτώσει, ξέρουν ε, ότι και ο τουρισμός συνδυάζεται με την αλία και ε, αλληλεπιδρούν. Βεβαίως υπάρχουν και πολλοί ε, διαφορετικές πραγματικότητες και διαφορές από περιφέρεια σε περιφέρεια με κάποια τροπολογία μπορεί να διαφωνήσουμε αν είναι ιδιαίτερα φωτογραφική για κάποια ιδιαίτερη περιφέρεια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ευρωπαϊκή υπόθεση. Μερικά πράγματα ανήκουν στην επικουρικότητα και θα πρέπει να αποφασίζονται επί τόπου. Αλλά ε, αυτός ο λευτικός τουρισμός μπορεί να λαμβάνει πολλές μορφές. Μας αρέσει πολύ η γνωμοδότηση και ευχαριστούμε για αυτή. Και σε γενικές γραμμές συμφωνούμε και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Εύανς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Ζήτη για ένα ενδιαφέρον ε, ζήτημα και στην Task Force για τον τουρισμό και σε αυτήν εδώ την Επιτροπή έχουμε εξετάσει τους τρόπους με τον οποίο μπορεί να συμβάλλει ένα τέτοιο είδους ε, αλευτικού τουρισμού στην ανάπτυξη των σχετικών κοινοτήτων και στη γενική ανάπτυξη αυτού του τομέα. Οπότε πραγματικά μιλάμε για μια πολύ σημαντική πτυχή και εγώ από την πλευρά μου έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες αλλά η δική μου πολιτική ομάδα υποστηρίζει αυτή την ε, ε, γνωμοδότηση. Εγώ εκπροσωπώ την Ουαλίου εμείς από την πλευρά μας οπότε έχουμε μια πάρα πολύ εκτενή ε, ακτογραμμή ε, πάρα πολλών μελίων, οπότε πραγματικά ε, θεωρούμε πως θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε περισσότερο τέτοιες δραστηριότητε σε συνεργασία και σε τέτοια σχέση με άλλες χώρες ειδικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί όπως είπε και ο συνάδελφος λίγο πιο πριν ο Κιθ Taylor, θέλουμε να επιτύχουμε την ενίσχυση των ε, συνεργειών μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμα και όταν το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν αυτό είναι, θα καταστεί ακόμα πιο σημαντικό για μας τις μικρότερες περιφέρειες, το να συνεργαζόμαστε δηλαδή εντατικότερα μεταξύ μας. Ε, ε, υποστηρίζω όλες τις βασικές τροπολογίες σε ό,τι αφορά την κοινή πρακτική, τις κοινέ σε marketing, την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών κονδολίων και επίσης ενημέρωση προς το ποιε είναι οι πηγές χρηματοδότηση και ποιο είναι ο τρόπο με τον οποίο έχουν αξιοποιηθεί διαφορετικέ χρηματοδοτήσει. Έχω επίση υποβάλει μία ε, ε, τροπολογία η οποία αναφέρεται ειδικότερα στο ζήτημα των γυναικών γιατί παραδοσιακά γίνεται αντιληπτό ο τομέα τη αλληλεία ω ε, ένα τομέα όπου τον κύριο λόγο, αν θέλετε, έχουν οι άντρε. Οπότε νομίζω πως θα πρέπει να εστιάσουμε λίγο περισσότερο στις τοπικές κοινότητες ε, και στο ρόλο που παίζουν εκεί, μπορούν να παίξουν εκεί οι γυναίκες και στο επίπεδο δηλαδή του αλευτικού τουρισμού. Κύριε Πέτρια Αγγενόβα, εκ μέρους της ε, DGMAR έχει το λόγο. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε και κύριε και κύριε Ευρωβουλευτές. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά για το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνει η Επιτροπή σας για τα ζητήματα αλληλείας, ειδικότερα ε, σε ό,τι αφορά τον αλληλευτικό τουρισμό. Εμείς εξετάζουμε αυτή την περίοδο ε, τις ε, τροπολογίες που έχουν υποβληθεί και αναμένουμε βέβαια και το, την οριστική έκθεση που θα θεωρηθεί του χρόνου. Και εκεί βέβαια εμείς θα οριστικοποιήσουμε από τη δική μας, από τη δική μας πλευρά τη δική μας έκθεση, αλλά μπορούμε να πούμε ότι κατά τη δική μας εκ πρώτης όψης ευθυγραμμίζονται οι περισσότερες τροπολογίες με την κατεύθυνση που ακολουθεί η Επιτροπή. Επίση, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για το γεγονό ότι έλαβε υπόψη του τι ε, τα επαγγελματικό ένα ζήτημα το οποίο είχαμε αναφέρει κατά τελευταία μα ε, συζήτηση και αναμένουμε με ενδιαφέρον την ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα κάνουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ο λόγο και πάλι τώρα στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω του συναδέλφου με τη σειρά μου για τι τροπολογίε του και όλα αυτά τα θετικά που προτείνουν. Προσπάθησα να τις λάβω όλες υπόψη μου. Μην νομίζετε ότι δεν μας ενδιαφέρει η θάλασσα εμάς και η αλία. Μας αφορά και το πρόβλημα και εμάς γιατί έχουμε αλία. Μπορεί να μην έχουμε θαλάσσες αλλά έχουμε λίμνες οι οποίες έχουν και ψάρια και ψαράδες. Και μέχρι τώρα ε, πραγματικά ξέρετε ότι αυτό ήταν αντικείμενο επιβουλών διαφόρων στο παρελθόν. Ολόκληρη πόλη έχουν γίνει για το ποιο ελέγχει τις λίμνες και τα ποτάμια. Ε, δεν είναι μόνο η θάλασσα. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο αλληλευτικός τουρισμός ε, αναψυχής ε, είναι πολύ ωραία τα ψάρια και του γλυκού νερού και των λιμνών και των θαλασσών μας και ελάτε να ψαρέψετε με το καλάμι σας στην Ουγγαρία. Παρακαλώ, μην το θεωρήσετε αγένεια. Αύριο έχω ένα πρόβλημα και δεν μπορώ να παρευρεθώ στην ψηφοφορία. Έχω μια ανελημμένη υποχρέωση. Θα πρέπει να πάω σε ένα διεθνές ε, συνέδριο στη Βρατισλάβα. Ε, και πρέπει να φύγω αμέσως. Παρακαλώ να μην με παρεξηγήσετε, δεν το κάνω από γένεια. Βεβαίως θα ε, παρακολουθώ τις εξελίξεις πολύ στενά. Ευχαριστώ πολύ. Και η πάνω στο Δούνευ είναι. Και χίλια χιλιόμετρα πιο κάτω ε, είναι εύξηνος πόντος, δεν είναι και τόσο μακριά από θάλασσα. Λοιπόν, <laughs> έχει την σημασία του αυτό. Αύριο ψηφίζουμε στην Επιτροπή Αλίας στις 10 Νοεμβρίου και στην Ολομέλεια θα πάει το Δεκέμβρη, φέτος ακόμα. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τριών λεπτών για τεχνικούς λόγους λέει. Τρία λεπτά διάλειμμα, παρακαλώ.

Θα ηρεγούμε πριν. Ναι, ναι,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 Να συνεχίσουμε τώρα. Τα τεχνικά προβλήματα λύθηκαν. Και τώρα προχωρούμε στις επενδύσεις, ανάπτυξη και τα κτλ. Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλων είναι μια έκθεση πρωτοβουλία τη Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη. Ο κ. Σουλτόφσκι είναι εισηγητή και έχει αμέσω το λόγο. Συνάδελφοι, καταρχά να ευχαριστήσω όλου του σκιώδει εισηγητές για τη δουλειά του και τη συνεργασία του για τι συμβολέ του. Δεν έχουμε δεν είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μα, όμω καταφέραμε να καταλήξουμε σε διάφορε τροπολογίε συμβιβαστικές. Και προσπάθησα να λάβω υπόψη μου όλες τις απόψεις, όλες τις τροπολογίες για να μην αγνοήσω κανενών στην τοποθέτηση. Βεβαίως θα ήθελα να σταθώ σε κάποιες όλους ιδιαιτέρως. Συμφωνούμε με το γεγονός ότι τα διευθυντικά ταμεία και τα επενδυτικά ταμεία μπορούν να μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε ένα ε, εύρωστο μεταφορικό σύστημα και δίκτυο στην Ευρώπη. Πρέπει να, θέτουμε, θέσουμε τις σωστές βάσεις για να προχωρήσει και το TNT, τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Πολλές από τις τροπολογίες λοιπόν επαναλαμβάνουν την ανάγκη καλύτερης χρήσης του ΕΦΣΙ, του Ταμείου των Στατικών Επενδύσεων, για τις ευρωπαϊκές μεταφορές, κυρίως τα αστικά κέντρα. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική διάσταση και θέλουμε να έχουμε αστικές μεταφορές που να λειτουργούν αποτελεσματικά αλλά και με χαμηλό κόστος. Αυτό είναι σημαντικό και για τα αστικά κέντρα τα ίδια, αλλά και για τη διασύνδεσή τους με τις γύρω περιοχές στις μεγάλες πόλεις. Ε, σημαντική λοιπόν εδώ η λειτουργία των διευθυντικών ταμείων. Άλλε τροπολογίε αφορούν το σωστό συνδυασμό μεταξύ κεντρικών αρχών και περιφερειακών αρχών για την σωστή κατεύθυνση των επενδύσεων. Από την οπτική γωνία των περιφερειών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ανάγκε του από την αρχή του σχεδιασμού. Οι ειδικότερε ανάγκε θα πρέπει να λαμβάνουν ειδική στήριξη με τη συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων τη Επιτροπή και του αναλόγου πόρου εφόσον χρειαστεί αυτό. Μια πραγματική τέτοια συνεισφορά μπορεί να επιτρέψει την ολοκλήρωση έργων και προγραμμάτων, ώστε να μην επιβαρύνονται περιτά οι Ένα θέμα που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλέ επίση, η ανάγκη η τωρινή χρηματοδότηση να διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα και στα πλαίσια των ερχόμενων πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών, ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν σωρευτικά όφελο από την ανανέωση του ευρωπαϊκού μεταφορικού δικτύου. Η Ανατολική Ευρώπη και η Κεντρική Ευρώπη περιλαμβάνει πολλέ περιφερειακέ περιοχέ, λιγότερο αναπτυγμένε οικονομικά και λόγω των ειδικών γεωγραφικών του ε, συνθήκων. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε τα επενδυτικά ταμεία και άλλου, είδου είδους τέτοια εργαλεία. Επίσης, η άμεση χρηματοδότηση για κάποια μεταφορικά δίκτυα, όπως και το κόστος οικοδόμησης υποδομών, πολλές φορές είναι ιδιαίτερα υψηλό και εκεί χρειάζεται μια ιδιαίτερη μερίμνα. Και τέλος, υπάρχει το θέμα της πρόσβασης στα διευθυντικά ταμεία και τα επενδυτικά ταμεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλές διοικητικές δυσκολίες Πολύ φραγμοί που δυσκολεύουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων σε αυτά τα ταμεία, σε αυτά τα κονδύλια. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε δική μέρη εδώ, ειδικά στην περίπτωση των μεταφορικών δικτύων. Το γραφειοκρατικό άχθο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που πρέπει να παλύψουμε για να πετύχουμε αυτόν το στόχο μα. Ε, με τη συνεργασία των σκιωδών εισηγητών, ελπίζω ότι αύριο θα μπορέσει η Επιτροπή μα να υπερψηφίσει τι τροπολογίε που ήταν το καρπό του έργου μα. Ευχαριστώ, Κάμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, εξ ονόματος της ομάδας μας και ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος της κυρίας Σουίτσα που ακόμα δεν έχει φτάσει. Ε, καταρχάς επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την ε, καταπληκτική και αγαστή συνεργασία για το θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Πάντα έχω την εντύπωση ότι στις μεταφορές Όταν μιλούμε για υποδομές και τα, τα, τα μία υποδομών θα πρέπει να παίξει περισσότερο ρόλο ο κλάδος των μεταφορών, θα πρέπει και ενδιαφερόμενοι να ε, το κυνηγήσουν. 13 είναι οι συμβιβαστικές ε, τροπολογίες που συζητήθηκαν και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα υποστηρίξει τις 12 από τις 13 αυτές. Μία τροπολογία, μάλλον δύο, των συναδέλφων σοσιαλιστών και δημοκρατών, της κυρίας Ζέντερ και της κυρίας Ριβόνταλόν, έχουν να κάνουν με την ενοχή των ε, εθνικών αρχών στις επενδύσεις ε, για τις μεταφορές. Δηλαδή ε, υπάρχει θέμα με το χρέος το κρατικό. Μα κοιτάξτε, ε, και σου λένε ότι όταν επενδύεις μεταφορές να μην προσμετράτε αυτό το χρέος. Εντάξει, αυτό μας φαίνεται ότι το παρακάνει λίγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ακούει τα πάντα ε, μπορεί να το συζητήσει με το Eurostat για το πώς καταγράφεται το χρέος και τι προσμετράτε εκεί. Ο Δήμος της Λιέγης ήθελε να κάνει πολλές επενδύσεις, αλλά δεν τον αφήσανε, διότι θα αυξανόταν το χρέος του Βελγίου. Ε, χρειάζεται λοιπόν ε, κάποια προσοχή αυτό. Είναι καλές οι τροπολογίες αυτές, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Ισμαήλ Ερτούκ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ στα αγγλικά ο κύριος Ερτούκ. Τώρα έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω τη θέση της Κριστίν Γοβόντα που είναι η σκιώδης μας συγγήτρια. Κριστίν, εν πάση την ξέρετε. Γοβόντα πώς τη λένε, ε, αυτό. Ε, δεν είναι εύκολο για βαβαρό, είναι λίγο γλωσσοδέτης αυτό το όνομα. Λοιπόν, να πω δύο λόγια από πλευρά της Κριστίνα Βονταλόν η έκθεση πηγαίνει σωστή κατεύθυνση και συμπεριλαμβάνει ε, διάφορα θετικά στοιχεία. Έξι-εφτά είναι τα σημεία που θα πρέπει αυτή τη στιγμή να κοιτάξουμε. Πρώτον, η ανάγκη να αυξηθεί στο μέγιστο η ε, συνεισφορά των διαρθρωτικών ταμείων για να επιτύχουμε τους στόχους ε, για την αστική ατζέντα και το θεματολόγιο για την κινητικότητα στις πόλεις. Επίσης, αν υπάρχει για περισσότερη συνέργεια για τα ευρωπαϊκά κονδύλια στον τομέα των μεταφορών. Έχει σημασία να ολοκληρωθούν τα σχέδια διασυνοριακών μεταφορών και να γίνουν οι συνδέσεις εκεί που λείπουν. Οι παραμεθόρες, επίσης, υπάρχει σημασία μεγάλη της εδαφικής και κοινωνικής συλλογής, η σύνδεση με τους στόχους των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, και να μειωθεί ο γραφειοκρατικός ε, φόρτος. Παρόλα αυτά, θέλουμε να τονίσουμε δύο σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπογραμμίσουμε ότι η μόχλευση των ε, χρηματοδοτικών μέσων παραμένει πολύ χαμηλή ε, και ε, στις μεταφορές. Οπότε η επιδοτήσει υποχορηγήσεις είναι ο καλύτερος τρόπος να επιδοτηθούν αυτά και όχι τα δάνεια και επίση θα πρέπει να ζητήσουμε μεγαλύτερη ευελιξία από τον προπολογισμό για να τονωθεί στα διευθυντικά ταμεία η κρατική συγχρηματοδότηση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η Επιτροπή μα να τοποθετηθεί για το θέμα αυτό, καθώ γνωρίζουμε όλοι ότι οι επενδύσει σε βιώσιμε υποδομέ μεταφορών χρειάζονται μεγάλη ε, κρατική παρέμβαση και δεν είναι αποδοτικέ τόσο πολύ ε, ε, για τον ιδιωτικό τομέα. Αυτά λέει η Κριστίν. Ευχαριστώ και τον Ισμαήλ και την Κριστίν ο Ντομινίκ Χικέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και για τη δουλειά του και για τη συνεργασία του. Θα στηρίξουμε όλες τις συμβαστικές από την ομάδα μου. Όμως, για κάποιες τροπολογίες, Πρόεδρε, μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές αποκλήσεις της απόψεις, ιδίω με αυτό που είπε και ο κ. Κάμπ, έχοντα υπόψη κάποιε γενικότερε σκέψει για την δημοσιονομική πολιτική των κρατών μελών και τι πολιτικέ διαστάσει που μπορεί να λαμβάνουν κάποια θέματα μεταφορών. Αυτό καλό είναι να το σκεφτούμε και ως προς την έκθεση και να μην προδικάσουμε κάποια ζητήματα λίγο περίπλοκα και ακαθόδη για κάποιους συγκεκριμένους τρόπους μεταφορών που μπορεί να προκαλέσουν ε, κάποιους ενδιασμούς. Στο σύνολό όμως στηρίζουμε τις συμβαστικές. Αυτό που ήθελα πάντως να επισημάνω προ την έκθεση και να προσθέσω είναι ότι ικανοποιηθήκαμε ιδιαίτερα που είδαμε ότι ο εισηγητής επιμένει στην ανάγκη να υπάρξει συνδυασμό των διαφόρων δημοσιονομικών ε, εργαλείων. Να υπάρξει αυτό το μίξ. Δηλαδή και τα περιφερειακά ταμεία και τα ειδικότερα και αυτά να συνδυαστούν με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία. Είναι πολύ σημαντικό και θα συνεχίσουμε να το επαναλαμβάνουμε. Αντιθέτω, θα ήθελα λίγο περισσότερο να τονιστεί κάτι που δεν έγινε, αν και υπόθηκε, είναι πόση σημασία έχει η καλή διαχείριση των ε, κονδυλίων με τον ε, πολιτή δημοσιονομικό ε, κανονισμό. Θα πρέπει να υπάρχει ένας δημοσιονομικός κανονισμός, δεν είναι βέβαια στόχος της έκθεσης αυτός και γι' αυτό δεν βάλαμε σχετική τροπολογία, όμως όπως ξέρετε ο δημοσιονομικός κανονισμό μπορεί να απαγορεύσει κάποια φορά τη χρήση των ε, σχετικών κομιλίων στι μεταφορέ. Αυτό θα πρέπει να το δούμε με του συναδέλφου τη Επιτροπή ε, Προπολογισμών και Ελέγχου των Προπολογισμών. Το τρίτο στοιχείο, κάτι στο οποίο επέμεινε πολύ συγκεκριτή και συμφωνούμε, είναι να ε, συνδυάσουμε τα εθνικά προγράμματα, αλλά να υπάρχει και εμβάθυνση της συνεργασίας των περιφερειακών με τα επενδυτικά ταμεία σε περιφερειακό επίπεδο και επίσης διασυνδέσεις διασυνοριακές. Και αυτό είναι ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση κάποιες ε, μικροαποκλήσεις ε, σε κάποιες επιμέρους ε, διατάξεις μπορεί να υπάρχουν, όμως στο σύνολο στηρίζουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ. αλλά δεν αναφέρθηκατε στο κενό των 800 μέτρων μεταξύ Βανεθάν και ε, Βρυξελών. Με εντυπωσιάζει αυτό. Ε, πάντως, ε, να δώσω τώρα το λόγο στην εκπρόσωπο της ε, Κάτρι Ούστολ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον εισηγητή. Ε, δεν θα μακρηγορήσουμε, γιατί δεν υπάρχει κάποιο σημείο από τον οποίο να διαφωνούμε. Ε, το σχέδιο δηλαδή της έκθεσης ε, και όλα τα σημεία που αναφέρει είναι πράγματι ευστοχά, αλλά θα ήθελα να τονίσω μια συγκεκριμένη πτυχή η οποία είναι σημαντική τόσο ε, τώρα όσο και για το μέλλον. Η σχετική λοιπόν έκθεση του 2016 της Επιτροπής αναφέρεται σε μια ανοιχτού τύπου πλατφόρμα δεδομένων και ε, εδώ βέβαια ενδιαφέρει πάρα πολλούς το από πού θα έρθει η σχετική χρηματοδότηση και έτσι λοιπόν εμείς εκ των προτέρων μπορούμε να πούμε όχι μόνο ανατομέα πού πηγαίνουν τα χρήματα αλλά μπορούμε να πούμε και συγκεκριμένα χιλιόμετρα οδών μεταφορών, για παράδειγμα δικών μεταφορών, ε, συνδεδομικών μεταφορών, ε, στα οποία κατευθύνονται αυτές οι επενδύσεις. Άρα λοιπόν έχουμε άνα κράτος μέλος, άνα περιοχή, άνα project, άνα πρόγραμμα, ποια είναι τα κονδύλια τα οποία έχουν, έχει υπάρξει δέσμευση, έχουν, έχει υπάρξει σχετική ε, ανάληψη αν θέλετε της δέσμευσης ούτως ώστε να επενδυθούν στο σχετικό τομέα των μεταφορών. Και αυτό νομίζω πως θα είναι πολύ σημαντικό για σας, ούτως ώστε να έχετε μία βάση, μία πλατφόρμα στην οποία μπορείτε να, να αναφέρεστε, ούτως ώστε όταν πλέον έρχεται σε επαφή με τους δικούς σας ε, πολίτες ε, να αναφέρεστε σε συγκεκριμένα στοιχεία. Ε, θα μπορείτε δηλαδή να βλέπετε με βάση αυτή την ε, ε, πλατφόρμα το πού βρίσκεται το κάθε έργο και σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Αύριο είναι η, στην, στην η συνεδρίαση, η ψηφοφορία, συγγνώμη, στη Ρέγγιο. Δεν θυμάμαι που Α, όχι, ο Κοσμάς Οτόφσκι καταρχήν ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω, όλα ήδη υπόθηκαν. Σήμερα... Όχι, αύριο, αύριο λοιπόν ψηφίζουμε εδώ. Πρόεδρος. Σα ευχαριστώ πάντω που τα είπατε κατευθείαν στα γερμανικά. Δεν χρειάζεται να βάλω τα ακουστικά μου. Λοιπόν, εμεί ψηφίζουμε αύριο η Ρέγγι ή τον Νοέμβριο. Μάλλον τον Νοέμβριο. Μάλλον τον Νοέμβριο θα ψηφίσει αυτή την έκθεση και μετά η Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο τη σήμερα σα διάταξη δηλαδή η ετήσια έκθεση σε ό,τι αφορά την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα σχέδιο νομοδότησης ε, ε, προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομικής Πολιτικής που είναι αρμόδια επί της ουσίας. Η Ζακλίν Φώστερ είναι η, αρμόδια συντάκτης. Ε, και ο Ζουλώση αναφέρει το γεγονό ότι δυστυχώ έχασε την πτήση τη και δεν μπορούσε να παρευρεθεί σήμερα εδώ. Θα κάνω εγώ την παρουσίαση τη συναδέλφου Φώστερ, ε, θα τη διαβάσω μάλλον στην αγγλική γλώσσα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ε, τοποθέτηση της η έκθεσή της υπογραμμίζει ε, τα κανονιστικού και άλλου ε, χαρακτήρα εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών που κατακαιρματίζουν την αγορά και δημιουργούν εμπόδια στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Άρα λοιπόν απαιτείται μεγαλύτερη πολιτική βούληση τόσο από την Επιτροπή όσο και από τα κράτη-μέλη προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά μεταφορών. Ένα, ένας ακόμα κεντρικός άξονας αυτής της ε, νομοδότησης είναι η πρόοδος που έχει εμπνευθεί, οι εξελίξεις στον τομέα των σχετικών τεχνολογιών και στον τομέα, στον κλάδο του τουρισμού. Ε, κατά την άποψη της συγκεντρίας, δεν θα πρέπει να γίνονται λεπτέ ω απειλή, αλλά ω ευκαιρίε για τη δημιουργία περισσότερου ανταγωνισμού, για τη δημιουργία ε, περισσότερων θέσεων εργασία και για κάτι το οποίο θα βελτιώσει σε τελική ανάλυση την κατάσταση των καταναλωτών. Επίση, καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την πρόθεση τη υπογραφή ε, συμφωνιών σε ό,τι αφορά τι εναέρειε μεταφορέ με ε, σημαντικέ σε τρίτε χώρε. Τέτοιου είδου μεταφορέ θα επιτρέψουν όχι μόνο καλύτερη πρόσβαση στην αγορά, αλλά θα παράσουν και νέε επιχειρησιακέ ευκαιρίε ε, στον ε, κλάδο αεροπορία Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντα έτσι θέσει εργασία και δημιουργώντα περισσότερο όφελο για του καταναλωτέ. Τέλο, η νομοδότηση αναφέρει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η ακαιρεότητα της ενιαίας αγοράς ώστε να υπάρχει θεμητή, θεμητός ε, και διαφανής ανταγωνισμός ε, μεταξύ των ε, διαφορετικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών και στον τομέα του τουρισμού. Σας ευχαριστώ πολύ, Λέω ο Πρόεδρο. Μα τα διαβάσατε πάρα πολύ ωραία στα αγγλικά, τα καταλάβαμε όλα. Μην παντεκράμπτε πάλι. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάλι εγώ είμαι. λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά και ε, ο συνάδελφος ε, Σαλίνη είναι καθοδόν. Όλοι καθοδόν είναι, έρχονται στις Βρυξέλλες. Ε, ο κύριος Σαλίνη λοιπόν έχει καθυστερήσει και αυτός να κάνω μερικά σχόλια εξ ονόματός του. Καταρχάς, ευχαριστεί την Τζάκη Φώσταρ και τον Τόμας Λοτόφσκι για ε, τη γνωμοδότηση αυτή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό που η Επιτροπή Μεταφορών γνωμοδοτεί ακριβώς για αυτό το θέμα και την έκθεση ανταγωνισμού της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, διότι είναι πολλά τα λεφτά για τις επενδύσεις. Έχουμε μεγάλη οικονομική δύναμη για να τονώσουμε τον ανταγωνισμό και ε, την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη και καλό είναι αυτό και καλό είναι που η Τζάκη Φώστερ κάνει αυτή τη γνωμοδότηση προς την ε, ΕΚΟΝ Υπάρχουν όμως μερικά σημεία που τον τελευταίο καιρό ε, απασχόλησαν την επικαιρότητα και αύριο θα ψηφίσουμε πρώτα απ' όλα τον κανονισμό για τις λιμενικές υπηρεσίες. Ο κανονισμός αυτός σε μεγάλο βαθμό θα ανοίξει περισσότερο την αγορά και πάντα γίνεται συζήτηση για το τι είναι ε, δημόσια υπηρεσία και τι είναι ιδιωτική, ας πούμε δημόσια παραμένουν οι πιλότοι, οι πλοηγοί. Ε, ε, άλλοι λένε ότι θα πρέπει τα ρεμολκά και οι πλοηγοί, οι πιλότοι να παραμένουν στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Εν πάση περιπτώσει είναι θέματα ανταγωνισμού και ανοίγει και αυξάνεται ο ανταγωνισμός και στον κλάδο αυτό. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει και το πακέτο για τις οδικές μεταφορές και το περιμένει και ο συνάδελφος Ισμαήλ Ερτούκ για θα το κάνει και η Επιτροπή μας. Ξέρουμε ότι οι οδικές μεταφορές ε, είναι ε, και ήταν ανέκαθεν πάρα πολύ ε, ανταγωνιστικές, αλλά όταν είσαι πάρα πολύ ανταγωνιστικός έχεις να κάνεις με καμποτάζ και με κοινωνικό dumping ή με ε, διάφορες, σε πάση περιπτώσει, ατασταλίες στις συνθήκες εργασίας των απασχολουμένων εκεί. Και αυτό έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό. Πέρυσι, την Άνοιξη, μάλλον φέτος την Άνοιξη, ολοκληρώσαμε το τέταρτο πακέτο για το σιδηρόδρομο και το τεχνικό σκέλος και το σκέλος της αγοράς. Για ορισμένους η αγορά δεν έχει ανοίξει αρκετά και αρχίζει γενομένης από σας γιατί εσείς την καταψηφίσατε πρόεδρε γιατί θεωρήσατε ότι δεν πηγαίνει αρκετά μακριά. Με εκπλήσει αυτό, είστε και πράσινος, αλλά όλοι έχουμε τις αδυναμίες μας, για να το πω έτσι, και τα αδύνατα σημεία μας. Ε, πάντως, ε, καλό είναι ε, που οι διασυνοριακοί περιορισμοί έρονται τώρα, ιδιαίτερα με τα τεχνικά ζητήματα του πακέτου και είναι καλό. Τέλος, Πρόεδρε, Σήμερα το μεσημέρι συζητούσαμε ε, για τα ευρωπαϊκά ταμεία και τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Από τη μια έχουμε τα διευθυντικά ταμεία και από την άλλη ε, το, την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, το ΣΕΦ και το ΕΦΣΙ, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Όλα αυτά είναι περισσότερες δυνατότητες για επενδύσεις ε, στις μεταφορές. Σε οικονομική βάση δεν θα πρέπει να φοβόμαστε τον ε, ανταγωνισμό, αλλά θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Ο συνάδελφος Σαλίνη επίσης αναφέρει κάτι για τις κρατικές ενισχύσεις. Είναι κάτι που ε, κρέμεται στα δαμόκλια σπάθη ακόμα και στην έκθεση αυτή και θα κάνει σχετικά τροπολογίες στην γνωμοδότηση της κυρίας Φώστερ. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Σαλίνη ε, θα τα βρει τελικά με την κυρία Φώστερ δεδομένου και της ε, πολιτικής έτσι, τοποθέτησης των δύο βουλευτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ισμαήλ Ερτούκ, στα αγγλικά. Να ζητήσω συγγνώμη γιατί οι σκιώδη μα κυρία Ταπαρντέλ δεν μπορούσε να είναι εδώ, οπότε να παρουσιάσω εγώ τι παρατηρήσει τη. Η σκιώδη των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στηρίζει το σημείο 4 για το όφελο του να εκμεταλλευτούμε τι ευκαιρίε που προσφέρουν οι ψηφιακέ τεχνολογίε. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιε στοιχεία στην έκθεση με τι οποίε διαφωνούμε. Συνολικά η εντύπωσή μα είναι ότι οι κοινωνικέ πτυχέ ε, σχεδόν δεν αναφέρονται καν, γιατί η ανταγωνιστικότητα σίγουρα στηρίζει την ανάπτυξη, όμω Ταυτόχρονα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει μια σωστή ολοκλήρωση τη ενιαία αγορά για τι μεταφορέ, χωρί να πληγούν τα κοινωνικά δικαιώματα όσων εργάζονται σε αυτόν τον τομέα, ούτε να υποβαθμιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, τα σημεία 1, 2 και 3 θα μπορούσαν να βελτιωθούν αν δοθεί περισσότερη έμφαση στην ανάγκη να βρεθεί το σωστό σημείο ισορροπία μεταξύ των ωφελών για τι επιχειρήσει και τι εταιρείε και την προστασία των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών. Ο τομέας των μεταφορών ως τώρα μας έχει προσφέρει άφθονα παραδείγματα για το πώς η ανοιχτή αγορά έχει οδηγήσει στην εκμετάλλευση των εργαζομένων. Ως προς το σημείο 2 συμφωνούμε με τον ισχυρισμό τη εισηγήτρια ότι πολλέ φορέ οι κανονισμοί για τι μεταφορέ δεν εφαρμόζονται σωστά. Και υπάρχει και μια διασύνδεση εδώ με το σημείο 7 τα μονομερή μέτρα που μπορεί να ε, υιοθετήσουν τα κρατημέλη. Από αυτήν την έννοια θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την ανάγκη για περισσότερο συντονισμό και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά προτίμηση με τη δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τι Οδικέ Μεταφορέ, που ψηφίστηκε από την πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών και με την αφορμή τη έκθεση για το κοινωνικό ντάμπινγκ. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Τρελέτκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι εγώ δεν αντικαθιστώ κανένα. Είμαι εγώ ίδιος και όδης Ω Ως προς το σχέδιο έκθεση είναι πολύ καλό το κείμενο. Ε, αυτό που εκτιμώ είναι ότι πραγματικά ε, επικεντρώνεται στο θέμα των μεταφορών. τραν trans-focused όπω τα έλεγα. Και δεν ε, μπαίνει καθόλου στο πεδίο των άλλων επιτροπών. Κατά δεύτερον, προσυπογράφω πλήρω σε αυτό που είπε η κυρία Φώστερ, ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης το κατά πόσο θα την εσωτερική αγορά των μεταφορών. Και πραγματικά οι δυσκολίες στην υλοποίηση της εφιστάμενης νομοθεσίας, εφόσον δεν είναι επαρκής, είναι σαφώς το βασικό πρόβλημα. Επίσης στηρίζομαι την ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στους ίσους κανόνες ανταγωνισμού μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, Παραδοσιακά ε, είναι κάτι που ισχύει αυτό και το έχουμε δει και στην περίπτωση νέων εταιριών και να τονίσω ότι ο δίκαιος ανταγωνισμός ε, είναι επιτακτική ανάγκη οπότε πρέπει να διακρίνω μεταξύ του προστατευτισμού και των ε, ισότιμων κανόνων ανταγωνισμού. Αυτό αναφέρεται στο σχέδιο του κειμένου όμως, γι' αυτό και μπορώ να συμφωνήσω. Και τέλος να πω ότι θα υποβάλω αρκετές τροπολογίες προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του δίκαιου ανταγωνισμού και της ε, ιδιαίτερης απόχρωσης που θέλουμε να έχει ως προς αυτό το θέμα το κείμενο και το είδαμε και στα πρόσφατα θέματα της συνεργατικής οικονομίας αλλά πραγματικά ήδη η γραμμή που έχει ακολουθήσει η κυρία Φώστερ είναι μια γραμμή στην οποία μπορώ σχεδόν πλήρως να προσυπογράψω. Ευχαριστούμε κυρία Κιλόνεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, μπόρεσα να έρθω στην ώρα μου, ίσως ε, χωρίς να μπορέσω να σας ευχαριστήσω αντικαθιστώντας κάποιον και θα μιλήσω φιλανδικό. Ε, το θέμα της εισηγήτριας, το θέμα που προσπαθήσει για να αναπτύξει το κείμενο, είναι ένα θέμα που διχάζει αρκετά τις πολιτικές ομάδες εδώ, όμως ο τρόπος που τα αντιμετωπίζει η κυρία Φώστερ είναι αρκετά επιτυχής. Μπορώ να συμφωνήσω στα περισσότερα τμήματα του σχεδίου κειμένου, διότι αφορούν τι διασυνοριακές μεταφορές και δραστηριότητες. Οι μεταφορές και ο τουρισμός, ε, η αεροπλοεία ε, αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό και σχέσεις ανταγωνισμού με τις τρίτες, προβλήματα στις σχέσεις ανταγωνισμού με τις τρίτες χώρες. Το Κοινοβούλιο λοιπόν πρέπει να τα διευθετήσει όσο μπορεί αυτά προστατεύοντας τις οδικές μεταφορές, τους εργαζομένους στον τομέα των μεταφορών και τονώνοντας τον ανταγωνισμό, ε, τον δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων χωρών. Υπάρχει και το πακέτο μέτρων για τις οδικές μεταφορές, ενώ στις σιδηροδρομικές μεταφορές παραδοσιακά η αγορά βασίστηκε σε εταιρείε που ήταν ε, ε, de facto μονοπόλια. Τώρα αυτό χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα για το πώς θα ιδιομορφωθούν τα πράγματα στο μέλλον. Εξαρθρώνεται το σύστημα με πρόσφατη νομοθεσία. Δεν ξέρουμε όμως τι επιπτώσεις θα υπάρξουν για τους ε, τελικούς καταναλωτές, τους επιβάτες και το σύστημα μεταφορών. Με την επανάσταση λόγω χάρη της ψηφιοποίησης. Οι εταιρείες πρέπει να μπορέσουν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και σε αυτό το τομέα. Ο ανταγωνισμό δεν μπορεί να είναι μια εύκολη συνταγή για την ευτυχία. Αλλά ούτε θέλουμε να γίνει και ο σίγουρο δρόμο ε, για τον άδη και την κόλαση. θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο νομοθετικό περιβάλλον σε αυτό το τομέα, ώστε να υπάρχει νομική βεβαιότητα, ασφάλεια και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορεί και δραστηριοποιούμενοι να ε, αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Ο τομέας των μεταφορών θα πρέπει ακριβώς αυτό να εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία των μεταφορών και τις ανάγκες των πελατών. Θα πρέπει λοιπόν οι κανόνες του παιχνιδιού σε αυτόν τον τομέα να έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Να ε, καλύπτουν τις ανάγκες του τελικού καταναλωτή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Τέιλορ. Άλλος ένας σκιώδης που είναι παρόν. Thanks, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τι κρίμα που δεν είναι εδώ η Τζάκη. Mm. Ελπίζω όμως ότι θα έρθει τις επόμενες φορές και πραγματικά ανυπομονώ να συνεργαστούμε για την έκθεση αυτή. Όπως είπατε, είμαι σκιώδης για τους πρασίνους. Είμαι πεπισμένος ότι ο μόνος τρόπος να πετύχουμε δίκαιο ανταγωνισμό και να δημιουργήσουμε ισότιμους κανόνες παιχνιδιού και ανταγωνισμού σε όλο το τομέα των μεταφορών είναι ε, αντιμετωπίζοντας το αληθινό κόστος του κάθε τρόπου μεταφοράς αντικειμενικά. Κοιτάξτε στην υποπαράγραφο 1, όπου λέει η Τζάκη ότι πρέπει να υπάρχει ανοιχτό και δίκαιος ανταγωνισμός λόγου χάρη. Νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, το κόστος του κάθε τρόπου μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τις ε, επιπτώσεις στην υγεία, τη ρήπανση, την ασφάλεια και τις κλιματικές αλλαγές. Διότι προς στιγμή αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν έχουμε τα επιθυμούμενα αποτελέσματα ούτε ισότιμους κανόνες παιχνιδιού, ούτε ανοιχτό και δίκαιο ανταγωνισμό. Οι πραγματικές τιμές, η δίκαιη φορολόγηση των μεταφορών και άλλα δημοσιονομικά μέτρα μπορούν να επιτρέψουν τη μετάβαση σε άλλους τρόπους, σε πιο βιώσιμους τρόπους μεταφορών, όπως τη εσωτερικής ναυσιπλοείας ή του συνδροδρόμου, καθώς και τις καλύτερες επιδόσεις του κάθε τρόπου, ως προς την αποτελεσματικότητα, το κλίμα και το περιβάλλον. Σκεφτείτε μόνο την αεροπλοεία, η αεροπλοεία και το τομέα των αερομεταφορών. παίρνουν πολύ μεγάλο ποσό έμεσων και άμεσων επιδοτήσεων στις πλάτες των ε, φορολογουμένων. Ε, έχουν πολλές εξαιρέσεις από φόρους και ΦΠΑ από τα κράτη κατά 43 δις ευρώ ετησίως περίπου για τα κάψιμα. Εδώ ε, τα κράτη-μέλη χάνουν πολλές πολύτιμες πηγές εισοδήματο χωρί να έχουμε πιο βιώσιμε μεταφορέ και τελικά καταλήγουμε να υπάρχει αθέμητο ανταγωνισμό. Όπω επίση πρέπει να θυμόμαστε και τη Συμφωνία των Παρισιών και τα ε, μέτρα υπέρ τη αναχέτηση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών. Έχουμε κάνει κάποια πρώτα βήματα, αλλά δειλά δεν έχουμε ακόμη λάβει δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών. Οι μεταφορέ θα πρέπει να φορολογούνται δίκαια ε, με δεσμευτικά και υποχρεωτικά μέτρα για τον έλεγχο τη αγορά. Όλε οι διεθνεί πτήσει από και προ την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εμπίπτουν στο ETS, το Σύστημα ανταλλαγή Δικαιωμάτων Μεταφορών εδώ θα φροντίσω να υποβάλω σχετικές τροπολογίες για να αντικατοπτριστούν σωστά οι απόψεις μας και οι ελλείψεις ε, της εσωτερικής και ε, διατροπικής ε, μεταφοράς του συνδυασμού των τρόπων μεταφοράς. Ανυπομονώ για τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με πολλά από όσα είπαν ήδη συνάδελφοι και έχει μεγάλη σημασία τα κοινωνικά ε, στοιχεία της ε, απασχόλησης να ληφθούν υπόψη και να μην έχουμε μια κούρσα ε, και ανταγωνισμό προς τα κάτω. Αυτό θα πρέπει να εκφράζεται με έντονο τρόπο στις ομοδοτήσει μας και ελπίζω να γίνει και με τις τροπολογίες. Τι λείπει όμως από αυτή τη νομοδότηση, η αναγνώριση των μεταφορών ως μια ζωτική σημασία σε υπηρεσία Δημόσια υπηρεσία. Πολλοί κόσμος είναι υποχρεωμένος να παίρνει ένα μέσο μεταφοράς για να πηγαίνει στη δουλειά του και να μην διχάσει. Ε, δεν είναι επιλογή του έχει κάνει μια εξαιρετική ε, μελέτη, υπηρεσία μελετών του Κοινοβουλίου και τη συζητούσαμε πέρσι, ε, που έχει να κάνει με την κοινωνική ένταξη και τις ε, δημόσιες μεταφορές και πώς συνδέονται αυτά τα δύο. Και θα πρέπει υπόψη μας να τα έχουμε στην πολιτική μεταφορών και να μην τα βάζουμε όλα στο τσουβάλι του ανταγωνισμού. Αυτό δεν ενισχύεται και από μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φετινή στις αρχές του έτους έγινε, για δημόσιες συμβάσεις και ε, μεταφορές που είδαν από το 2008 που ξέσπασε η κρίση η χρηματοπιστωτική υπήρξαν μεγάλα προβλήματα σε πολλά κράτη-μέλη ακριβώς διότι οι δημόσιες μεταφορές δεν στηρίχθηκαν ε, επαρκώς. Και αυτό ε, είναι μια πολύ ωραία ομαλή μετάβαση στο επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε αλλά δεν ε, διαφωνώ καθόλου με τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση και χαίρομαι για τη σημερινή συζήτηση, αλλά χρειάζεται ε, σημαντική βελτίωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίλσον. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα απ' όλα ε, στα κοινωνικά ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά και έχουμε κατά πλειοψηφία λάβει μια ε, απόφαση για το κοινωνικό ντάμπινγκ και ξέρουμε ποια είναι η άποψη της πλειοψηφίας. Αυτό θα επηρεάσει και το κείμενό μας. Άλλη παρατήρηση. Μιλήσαμε για τη βελτιστοποίηση ε, της αξιοποίησης των ταμείων επενδύσεων. Maximizing το λένε αυτό στα αγγλικά. Δηλαδή, μεγιστοποίηση, όχι μόνο βελτιστοποίηση. Εγώ μιλώ για τη χώρα μου, αλλά και σε άλλες χώρες τι έχουμε διαπιστώσει. Ότι όταν έχεις ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό, ε, είναι σημαντικές οι επενδύσεις, ε, γιατί έτσι αναπτύσσεται ο τουρισμός. Επίσης, προσπαθήσαμε να αντλήσουμε κονδύλια ε, για τη χρηματοδότηση τέτοιων υποδομών δεν μπορούν τα περιφερειακά ταμεία και το Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων να επενδύσουν για το ίδιο έργο. Δεν επιτρέπεται δηλαδή. Δεν μπορεί να έχει διασταυρούμενη ε, χρηματοδότηση. Μα αυτό είναι βελτιστοποίηση και μεγιστοποίηση της εισφοράς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάτι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να συνενωθούν όλες οι δυνάμεις και να επενδυθούν τα απαραίτητα κονδύλια σε ένα στρατηγική σημασίας έργο. Αυτό θα σας προτείνω σε σχετική τροπολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω γράψει και τον εαυτό μου τώρα στον κατάλογο. 12 χρόνια είμαι μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όταν συζητούμε αρχές, η αρχή ο χρήστης πληρώνει, η εσωτερήκευση ε, του εξωτερικού κόστους και ο ρηπαίνων πληρώνει, όλοι συμφωνούμε διακομματικά, διακρατικά, θαυμάσια ομόνια και συναντήληψη. Όταν όμως πρόκειται για τις μεταφορές, και έχουμε ένα συντηρητικό βουλευτή Γερμανό που το είπε, ε, ότι στις μεταφορές η οικονομία της αγοράς έχει εξουδετερωθεί και αυτό μας εμποδίζει. Μα αν δούμε ποια είναι τα μέσα μεταφορών ε, που βλάπτουν το κλίμα, έχουν, ε, το κλίμα, έχουν εξαιρετικές ευνοϊκές ρυθμίσεις και οικονομικές και πολιτική στήριξη, ενώ εκείνες που είναι φιλικοί προς το περιβάλλον και εκείνα τα μέσα μεταφορών έχουν ε, πολύ δυσμενή μεταχείριση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εκείνα ε, κοιτάει μόνο τις οδικές μεταφορές, το σιδηρόδρομο, τις πλωτές οδούς, την αεροπορία και εκεί θα πρέπει να είναι όλα εντάξει. αν συγκρίνουμε όμως τους τομείς, ε, δεν έχει ε, κανένα ρόλο να παίξει. Ξέρετε το προσφυλές μου θέμα, 30 δισεκατομμύρια ε, χαρίζουν στις αεροπορικές εταιρείες κάθε χρόνο οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι γιατί δεν πληρώνουν φόρο για την κυροζήνη ενώ οι άλλοι να πληρώνουν ο χρήστη του σιδηροδρόμου κτλ. Γι' αυτό είναι τόσο φθηνές οι πτήσεις και είναι και εχθρικέ προ το περιβάλλον. Και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Μα τι στο καλό κάνετε εκεί πέρα. Έχει μαλλιά σε γλώσσα μου να τα λέω. Τι κάνετε, ε, πώ φροντίζετε οι αρχέ αυτέ για τι οποίε συμφωνούμε να εφαρμοστούν και στι μεταφορέ. Και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να δώσω το λόγο στον κύριο Στέφαν Ζήμων από την Αρμόδια Γενική Διεύθυνση για να μα διαφωτίσει. Παρακαλώ. Τρεις έχουμε από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και εμεί πρόχνεστε. Δεν πειράζει, περιμένουμε. Γιατί το περιεχόμενο ουσία έχει νόημα και όχι ταχύτητα. This question not seem in the για τον ανταγωνισμό. Εδώ φαίνεται να υπονοείται τις άμεσες επιδοτήσεις που θα μπορούσαν να είναι παράνομες, τις κρατικές επιδοτήσεις. Αυτό τώρα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σε κάποιες περιοχές βέβαια έχουμε κοιτάξει να πατάξουμε την ε, φοροαποφυγή, αλλά σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα είναι νομοθεσία των κρατών μελών αυτή και δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Δεν έχουμε αναλάβει δράση σε αυτό το τομέα. Μου επιτρέπετε σύντομα να πω κάτι ε, σε σχέση με αυτό. Στη Γερμανία πώς έχουν τα πράγματα. Από τα 23 αεροδρόμια, τα 17 είναι λιματικά που παραμένουν στη ζωή γιατί κατά κάποιο τρόπο παίρνουν κρατικές ενισχύσεις. Αλλά όταν ε, είχαμε ε, ε, ε, Βερολίνο ε, Βρότσλαβ, ένα, μια γραμμή σιδηροδρομική, καταργήθηκε το δρομολόγιο γιατί λέει ήταν ασύμφορο και δεν μπορούσαμε να δώσουμε κρατική ενίσχυση. Δεν είναι μόνο φορολογική. Ξέρω ότι έχετε επέμβει για κάποια αεροδρόμια, το Χάν τους δύο γέφυρες της Φαϊμπρούκεν, αλλά για άλλα όχι και γιατί οι κρατικές ενισχύσεις γίνονται δεκτές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους μεν, αλλά για τους δε όχι. Αναφερθήκατε στο πρόβλημα των, των και των σχετικών συνδέσεων. Ο, ε, η σχετική αγορά από την δεκαετία του 1990 είναι απελευθερωμένη. Ε, ε, για πολύ καιρό δηλαδή αναφερόμασταν στους αερολιμένε ως υποδομή, αλλά μετά από την απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση Χάλε Λάιψιχ, αποκρισταλώθηκε τελικά η άποψη, αν θέλετε, ότι μπορεί να υπάρξει κρατική ενίσχυση απέναντι σε τέτοιου είδους υποδομές ε, για τους αερολιμένες. Ε, εμείς αντιδράσαμε σε αυτό. Ε, το 2014 υιοθετήσαμε τις σχετικές κατευθυντηρίες γραμμές για τους αερολιμένους και ξεκινήσαμε, ε, ανοίξαμε μια σειρά από διαφορετικές ε, υποθέσεις, ε, διαδικασίες σε μια σειρά από κράτη-μέλη και πραγματικά γνωρίζω ότι και στη Γερμανία μόνο τρεις αερολιμένες πραγματικά κερδίζουν χρήματα, δηλαδή δεν έχουν λύματα και έχουμε βέβαια θέσει και μια σχετική προθεσμία η οποία τρέχει ακόμα για κάποια χρόνια όπου επιτρέπονται κάποιες ενισχύσεις. Οπότε σας ζητώ να μας δώσετε λίγο παραπάνω χρόνο γιατί υπάρχει αυτή η προθεσμία. Ε, κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει έγκυρα η σχετική διαδικασία και γι' αυτό υπάρχουν αυτές τις καθυστερήσεις. Ο Ναι, Πρόεδρε. Πρόεδρε, για να καταλάβω λίγο. Πολύ ωραία που απαντήθηκαν οι δικές σας ερωτήσεις, αλλά Θέλουμε και άλλα σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κείμενο της Ζάκη Φώστερ, έτσι δεν είναι. Γίνεται αυτό, έτσι, εμπαρόδο, ξέρω εγώ. Also ich kann... Ο πρόεδρος, εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σίγουρα. Ich weiß jetzt, von Ihnen... Δεν ξέρω ποιο έχει σειρά από εσά, αλλά με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουμε να ακούσουμε τη θέση σα για το κείμενο, αλλά και για τη συζήτηση εδώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Okay, I'm DG Competition and not the Commission, but at least from the... Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Ε, οπότε ως ε, DG Competition θα σας απαντήσω. Εμείς ε, συμφωνούμε με τα όσα αναφέρει, δηλαδή και εμείς καλούμε την Επιτροπή να επιταχύνει την υιοθέτηση του τέταρτου πακέτου για τους σιδηροδρόμους, δηλαδή πράγματι να υπάρξει, θα πρέπει να υπάρξει πίεση απέναντι και στα κρατημέλα αλλά και στο Κοινοβούλιο τους ώστε να υιοθετήσουν και να εγκρίνουν τη σωστή νομοθεσία. Μετά από την Επιτροπή ο Κοσμάς Λατόφξη έχει και πάλι το λόγο εξ ονόματος της συναδέλφου Σαγκρίν Φώστερ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα τα σχόλια που κάνατε. Σας ευχαριστώ εξ ονόματος της συναδέλφου Φώστερ και ε, αναμένω κι εγώ με ενδιαφέρον την ε, περαιτέρω συζήτηση που θα κάνουμε για αυτό το ζήτημα. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 13 Οκτωβρίου. Η ψηφοφορία στην Τραν είναι στις 10 Νοεμβρίου, η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΚΟΝ 5 Δεκεμβρίου και στην Ολομέλεια η ψηφοφορία δεν γνωρίζουμε ακόμα την ημερομηνία για την ψηφοφορία. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη, στο επόμενο σημείο της μέσης σας διάταξης, δηλαδή ε, την ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με ε, συντάκτη της Μοδότης τον Σλαβίλου Μπεράτσι, ο οποίος δεν παρευρίσκεται σήμερα εδώ και έχουμε συνηθίσει πια να απουσιάζουν, αλλά η Λούση Άντερσον θα τον εκπροσωπήσει, οπότε της δίνουμε κατευθείαν τον λόγο. ναι, ε, χαίρομαι για το γεγονό ότι μου ζήτησε ο Μπογκούσλαβ να τον αντικαταστήσω σε ό,τι αφορά την παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότηση του, σε ό,τι αφορά την έκθεση σχετικά με τι γραμ... χρηματοδοτικέ δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πάντοτε συνέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό στα έργα ε, υποδομών ε, μεταφορών που βέβαια συμβάνουν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη, του ρυθμού ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το γνωρίζω πολύ καλά και από τι επενδύσει ε, στη δική μου χώρα και στο Λονδίνο. Ε, πέρα τώρα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπάρχουν και άλλε πηγέ χρηματοδότηση των έργων μεταφορών, όπω για παράδειγμα η η διευκόλυνση ε, για την Ευρώπη, τα διαθροτικά ταμεία και ό,τι καθεξής. Άρα είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρξει ένας ε, συντονισμός μεταξύ των διαφόρων αρχών χρηματοδότησης και πηγών χρηματοδότησης, δηλαδή μεταξύ των κρατών μελών της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των άλλων αρχών. Και σύμφωνα με τον Μπόγκουσλαβ θα πρέπει αυτός ο συντονισμός να γίνει με βάση τα όσα προβλέπει ο κανονισμός για τα ευρωπαϊκά δίκτυα της μεταφορών. Δηλαδή. Επίσης το Ταμείο για τα Διευθυντικά Ταμεία, από την πλευρά του εστιάζουν σε κάποια έργα, σε κάποια συγκεκριμένα project, τα οποία δεν είναι τόσο ελκυστικά για του ιδιωτικού επενδυτέ, ενώ ε, από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπάρχουν ε, τέτοια ε, project, τα οποία μπορούν να κινητοποιήσουν ακριβώ περισσότερο το ιδιωτικό κεφάλαιο. Γι' αυτό το λόγο, η συγκητή σε αυτό το σχέδιο τη γνωμοδότησή του ε, προτρέπει να υπάρξει περισσότερη αλληλοσυμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφορετικών πηγών χρηματοδότηση. Ο ε, συντάξει νομοδότη επίση ε, τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην γεωγραφική ισορροπία των επενδύσεων που γίνονται με τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα πρέπει δηλαδή να ληφθεί περισσότερο υπόψη περιφερειακή διάσταση και θα πρέπει να υπάρξουν κατευθυντήριε γραμμέ για τι εταιρικέ σχέσει ιδιωτικού δημοσίου τομέα, ώστε να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία ε, για τον τον έργων ε, που χρηματοδοτούνται από την ε, Τράπεζα Επενδύσεων. Με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, θα αποφευχθούν και παραβάσει οι οποίε απλά βασίζονται στη διαφορετική ερμηνεία των σχετικών κανόνων. Επίση, ο κύριος Λιμπεράση τάσεται υπέρ της παράτασης της των σχετικών επενδυτικών και ελευθερικών ταμείων στο 2000, ε, ε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τη σχετική πολιτική στο 2030. Βιμ, πάλι εσύ είσαι. Ε, ξέρετε, έχουμε διάφορα προβλήματα. Δευτέρα απόγευμα, ο καθένας ταξιδεύει. Ε, έχουν άλλες δραστηριότητε οι άνθρωποι. Καταρχάς, λοιπόν, θα ήθελα να απευθυνθώ στον εισηγητή τον κύριο Λιπεράτσκι και την κυρία Άντερσον κατ' επέκταση και να τους ευχαριστήσω. Είναι πάρα πολύ διαφωτιστική αυτή η γνωμοδότησή τους. Πρόκειται για μια ετήσια έκθεση, όπως γνωρίζουμε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά και με βάση τα όσα λέει ο κύριος Λιμπεράτσκι, είναι αλληλένδετα τα θέματα μεταξύ τους. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι μια πολύ μεγάλη τράπεζα που επενδύει πολύ στις μεταφορές. Λέει ο κύριος Λιμπεράσχη ότι 14 δισεκατομμύρια ευρώ παρακαλώ πέρυσι, τα τελευταία χρόνια μάλλον, έχουμε αντλήσει για τον κλάδο των μεταφορών από την ΕΤΕΠ. Αυτό είναι πραγματικά ε, σεβαστό ποσό. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, συνεπώς, όμως υπολείπεται. Αλλά αν δείτε και διαβάσετε τι χρηματοδοτεί και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επιδήσεων και ποια είναι αυτά τα έργα. Καταλαβαίνετε ότι είναι έργα υποδομής που χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλο χρόνο για την προετοιμασία. Και ό,τι έχουμε κάνει το 2015 η επενδύση δεν αποδίδει ε, το 2016, φτάνει μέχρι το 2018, ίσως και πιο μακράς πρωίς να είναι. Άρα θα ήταν ενδεχομένω καλό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προσέχει λίγο περισσότερο αυτά τα θέματα και να δίνει μεγαλύτερη δημοσιότητα και διαφήμιση. Ότι και με το ΕΦΣΙ, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, επενδύει στις μεταφορές, γιατί ακούω διάφορα πράγματα και ψιθύρους και θορύβους, ότι τα πράγματα πάνε καλά με το ΕΦΣΙ, αλλά πούντα. Δεν τα έχουμε δει ακόμα. Μετά, επενδύσεις στις βιώσιμε μεταφορές Είχαμε την COP21 και επίκειται τώρα η συμφωνία του ΑΙΚΑΟ. Ε, βλέπει να κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα. Ε, αηφορία, καινοτομία, συχνά είναι συνδεδεμένα αυτά και βιωσιμότητα και έχει μεγάλο ρόλο να διαδραματίσει και μπορεί η ετέπεκη. Και τέλος, η εξάρτηση από τις κρατικές ενισχύσεις εδώ μέσα το λέμε και blending αυτό καμιά φορά, θα πρέπει να διδαχθούμε ε, να συνδυάζουμε διάφορους τρόπους επενδύσεων που μπορεί να είναι και δάνεια και ε, grants, επιδοτήσεις δηλαδή που δεν επιστρέφονται. Και σε πολλά κράτη, ε, αυτοί που ασχολούνται με την ανάπτυξη και την, το σχεδιασμό των προγραμμάτων και των έργων, δεν το ξέρουν. Ε, δεν, δεν ξέρουν πώς να το χρησιμοποιούν. Και στην έκθεση Λιβεράτσικη λοιπόν αναφέρουμε αυτό το blending, να υπάρχει ένα χαρμάνι διαφόρων ε, μορφών χρηματοδότησης. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Ρικέ. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω όσα υπόθηκαν. Θα πρέπει να κοιτάξουμε να μελετήσουμε σωστά τα θέματα της έκθεσης, να τονίσω από αυτά που υπόθηκαν ότι η ΕΤΕ είναι βασικά τράπεζα. Ο τρόπος που λειτουργεί η ΕΤΕ, παρόλο που είναι μια δομή της Ένωσης, δεν έχει να κάνει με τα πολιτικά θεσμικά όργανα της Ένωσης. Και αυτό σωστά τονίστηκε. Υπάρχει πολλή δουλειά από την πλευρά της ΕΤΕ για τη διάρθρωση Τη δουλειά αυτή με του κρατικούς φορεί των κρατών μελών και των περιφερειακών εκπροσώπων των κρατών και τι οικονομικέ του δραστηριότητε. Από αυτήν την σκοπιά τονίστηκε ότι έχει πολύ σημαντική δουλειά να κάνει η τράπεζα. Οι αρχές των επενδύσεων, οι, αρχές της, οι επενδύσεις στις υποδομές είναι προφανώς αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Όμως, κάτι που είναι και επικαιρό, δεν υπάρχει δομική διάρθρωση μεταξύ των οργάνων της Επιτροπής που ασχολούνται ε, οργανικά με την ε, χρηματοδότηση και της ΕΤΕΠ. Είναι διαχωρισμένε οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολούνται με την χρήση των ε, διευθυντικών ταμείων, των ειδικών ε, ταμείων όπω το ε, Διευκόλυνση Διασύνδεση τη Ευρώπη και δεν συναρθρώνονται αναγκαστικά ούτε με την ΕΤΕ ούτε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ο μηχανισμός εγγύησεων που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά ελέγχεται πλήρω από το Διοικητικό Συμβούλιο τη Τράπεζα. Του μετόχου τη Τράπεζα. Δεν. Ε, ε, εδώ λοιπόν είναι θέμα σωστής συνδιάρθρωσης των ε, διαφόρων φορέων μεταξύ τους. Και ως προς το ετήσιο, την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της τράπεζας, Πρέπει να δούμε τη διασύνδεση των πολιτικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ΕΤΕ. Γιατί υπάρχει ο μηχανισμός των εγγύσεων, αλλά υπάρχει και η έλλειψη του σωστής ε, του σωστού κρίκου που θα συνδέσει τα δύο μεταξύ τους. Κατά τα άλλα ισχύουν οι κλασικές παρατηρήσεις που κάνουμε ως συνήθως για την λειτουργία της τράπεζας. Αλλά καλό θα ήταν να μελετήσουμε και τα ειδικότερα θέματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κίλωνεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, τον κύριο Λιμπεράτσκι, για την εξαιρετική του αυτή εργασία. Θα ήθελα να θυμίσω ότι μπορεί να το έχουμε ξεχάσει, γι' αυτό το θυμίζω. Την περασμένη εβδομάδα ε, υπερψηφίσαμε τη Συμφωνία του Παρισιού κατά της κλιματικής αλλαγής η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν θα σταματήσει επειδή έκανε πανηγυρική συνεδρίαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που χρειάζονται είναι συγκεκριμένα μέτρα, άρα και χρηματοδότηση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε <coughs> λοιπόν, διότι ε, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να μειώσουμε την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, να έχουμε καθαρές μορφές ενέργειας και έτσι να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και στις μεταφορές φυσικά. Θα πρέπει ε, να μιλήσουμε συνολικά για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και θα πρέπει να το δει και η Επιτροπή μας ας πούμε, η αναθεώρηση των μεθόδων, η συγκρισιμότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούμε, έτσι ώστε να μπορούμε να μετράμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων των έργων, με τρόπο πολύ πιο συγκεκριμένο και ορατό. Άλλη παρατήρηση. Ε, θα επιθυμούσα να αλλάξουμε νοοτροπία. Να μην μιλάμε για υποδομές μεταφορών ως μοναδική λύση, αλλά να μάθουμε να βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα γενικότερα στις υποδομές, τις υπηρεσίες μεταφορών και τις λειτουργίες των μεταφορών. Για παράδειγμα, παράδειγμα αυτοματοποίηση των υπηρεσιών μεταφορών. Αυτό ε, αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, πάρα πολύ ε, ταχύς. Σήμερα επενδύουμε με λάθος τρόπο, γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη οι επενδύσεις αυτές τα νέα είδη χρήσης των μεταφορών και αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις. Εγώ δεν θα μιλούσα μόνο για υποδομές μεταφορών, αλλά για υπηρεσίες μεταφορών. Και θα κάνουμε αντίστοιχη τροπολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ρόμπερτ Ζήλε. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα, αλλά να ευχαριστήσω τον κύριο Λιμπεράτη για την έκθεσή του. Ε, η έκθεση αυτή για το πρώτο τμήμα λειτουργίας της ΕΤΕ είναι περίπου αυτό που είχαμε προβλέψει και από την Επιτροπή μας. 50% των επενδύσεων αυτών κατευθύνθηκαν προς τα λεγόμενα παλιά κράτη-μέλη. Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης δεν ωφελήθηκαν. Δεν χρηματοδοτήθηκε κανένα σοβαρό έργο εκεί. Υπάρχει σαφής έλλειψη ισορροπίας λοιπόν, η οποία θα ενταθεί με το καιρό. Εάν κοιτάξουμε τι είχε προγραμματιστεί, τα ποσοστά γεωγραφικής συγκέντρωσης ε, ήταν περίπου στα 45% με τις αρχικές προβλέψεις. Η ισορροπία όμως αυτή δεν επετεύχθη. Τρεις μεγάλες χώρες αποφελούνται. Και αν μάλιστα δούμε και τον τομέα της ενέργειας σε συνδυασμό, όπου 30% είχε προβλεφθεί για υποδομές και έργα σχετικά με την ενέργεια, εκεί πήγαν και τα περισσότερα κονδύλια. Τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί και αντιμετωπιστεί εκ των προτέρων. Υπάρχει τεράστια έλλειψη ισορροπία. Στην ε, συνάντηση στην Πρατισλάβα αποφασίστηκε το ΕΦΣΥ να, να παραταθεί στη λειτουργία του για μια διετία. Αλλά τι θα αλλάξει με αυτό. Πραγματικά είμαι ιδιαίτερα επικριτικός ως προς τα όσα συμβαίνουν εργαστήκαμε για να αναπτύξουμε μια σωστή πολιτική μεταφορών και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τρόπους μεταφορών περιβαλλοντικά φιλικούς, όπως του σιδηροδρόμους, τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Βλέπουμε όμως η χρηματοδότηση να πηγαίνει αλλού. Ουσιαστικά κατευθύνεται στους τρόπους μεταφορών, όπου μπορεί κανείς εύκολα και γρήγορα τελικά να έχει οικονομικό κέρδος. Πιστεύω λοιπόν ότι μέσω της έκθεσης Λιμπεράσκη θα μπορούσαμε, θα μπορούσαμε τουλάχιστον να επιχειρήσουμε να τα επισημάνουμε αυτά τα προβλήματα και κατά πάσα πιθανότητα αν μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτήν την πολιτική τάση σε όλες τις πολιτικές της εκφράσεις. Δηλαδή από το πώς οι μεταφορές επιτυγχάνουν τους μακροπρόθεσμους στόχους και ο κύριος Κόνερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, ο Χέλαντ Ρόιτερ βρίσκεται εδώ μαζί μα, οπότε θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε τα όσα έχει να μα πει, παρότι δεν παρεμπρέθηκε στη συζήτηση εδώ. Αλλά βέβαια έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, οπότε ελπίζω πω θα μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα, το ότι δεν ήταν εδώ δηλαδή κάτι στη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους τους παρευρισκόμενους ε, βουλευτές. Ε, πράγματι δεν ε, άκουσα τη συζήτηση, οπότε είναι λίγο δύσκολο να δώσω απαντήσεις άμεσα όσους πήραν το λόγο. Εκείνο όμως που θα ήθελα να πω από τη δική μας πλευρά είναι ότι αυτό που είδαμε κατά τελευταία δύο χρόνια είναι πως η διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη αναπτύσσεται με πολύ θετικό τρόπο. Γνωρίζετε πως το σύνολο δηλαδή των κοντιλίων που είχαν δεσμευτεί έχουν απορροφηθεί γύρω στα 70 δις δηλαδή. Έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλες τις την εκδήλωση ενδιαφέροντος ε, και έχουμε μία σειρά από έργα τα οποία μπορούμε να προωθήσουμε και να επιλέξουμε ε, στην, ε, σε μελλοντικέ προκήρυξει για την εκδήλωση ενδιαφέροντο, εάν πράγματι εγκριθεί περαιτέρω χρηματοδότηση. Σε ό,τι αφορά το ΣΕΠ, προφανώ εδώ εστιάζουμε σε περισσότερη προστιθέμενη αξία διασυνοριακά και ειδικότερα σε ό,τι αφορά φιλικέ προ το περιβάλλον φιλικού προ το περιβάλλον ε, τρόπου μεταφορών και βέβαια πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη την ε, περιφερειακή ισορροπία. Ε, τώρα, έχουμε δει ε, μία σειρά από project τα οποία εστιάζουν στο rolling stock of shipping στο τροχείο υλικών και από εκεί και μετά έχουμε δύο ακόμα εγκεκριμένα green shipping schemes σε ύψος 3,5 δισεκατομμυρίων, δηλαδή συνολικό ύψος αυτών των προγραμμάτων βρίσκεται στο 12, στα 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτή η επιτυχία του ΕΦΣΙ οδήγησε ε, την Επιτροπή στο να διπλωσιάσει τη δική της ε, πρόταση ε, και σε ό,τι αφορά το, τη χρονική περίοδο όσο και σε ό,τι αφορά ε, τα κονδύλια, δηλαδή να προσθέσει άλλα 500 εκατομμύρια ευρώ στη χρηματοδότηση και να πάει το πρόγραμμα έως το 2020 ώστε να μπορέσουμε να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο στα φιλικά προς το περιβάλλον έργα και προκειμένου να λάβουμε ακόμα καλύτερα υπόψη μας αυτή την αρχή της συμπληρωματικότητας και εστιάζοντας και σε διασυνοριακά έργα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πολύ θετικές εξελίξεις και η έκθεση που συντάσσει η δική σας Επιτροπή συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν άκουσα λοιπόν τη συζήτηση, Πρόεδρε, και κατά συνέπεια θα είμαι σύντομος, θα σταματήσω εδώ και βέβαια είμαι στη διάθεσή σας για να δώσω απαντήσεις και από εκεί και μετά στην συνάντηση που θα ακολουθήσει θα είμαι στη διάθεσή σας. Η Λούση Άντερσον έχει παντού. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα ενημερώσω τον κύριο Λιμπεράσχη και επειδή δεν άκουσα εκείνο τη συζήτηση, θα φροντίσω εγώ να ανακεφαλαιώσω όσα υπόθηκαν. Οι βασικέ παρατηρήσει που έτειναν να κάνουν οι περισσότεροι συνάδελφοι και επειδή υπάρχει μια σχετική συνένεση στα περισσότερα θέματα, όσα έχουν να κάνουν με τον υπάρχει καλύτερη ανάμειξη των δημοσιονομικών εργαλείων για την επίτευξη και την ολοκλήρωση έργων, η δημιουργική χρήση των διαφόρων πηγών, όλα αυτά ακούστηκαν από πολλού. Η φύση τη λειτουργία τη ΕΤΕ είναι τράπεζα, σωστά υπόθηκε και αυτό και γύρει άλλες βασικές κατευθύνσεις για την έκθεση. Οι περισσότεροι πραγματικά ε, εκφράστηκαν υπέρ της ανάγκης γεωγραφικής ισορροπίας μεταξύ παλιών και νέων κρατών μελών, σημαντικό στοιχείο και βεβαίως και η περιβαλλοντική διάσταση. Πολλά θέλουμε να κάνουμε και άλλα πρέπει να βεβαιωνόμαστε τουλάχιστον τα έργα και τα προγράμματα ε, ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε η περιβαλλοντική φιλικότητά τους να είναι ένα από τα πρωταρχικά τους στοιχεία. Επίση, ο συντονισμό είναι καθοριστική σημασία. Ο συντονισμό, όπω είπε και ο Μπόγκο, λάβει συμπληρωματικότητα και η προσθετικότητα τη χρηματοδότηση. Άρα, νομίζω ότι γενικώ υπάρχει ευρεία σύμπνοια για την έκθεση αυτή και του στόχου τη. Ξαναζήτησε το λόγο ο κύριο Ρόιτερ. Συμφωνούμε να το, το ξαναδώσουμε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Ναι, θα ήθελα να απαντήσω λίγο σε ένα συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με αυτό που είπατε τώρα ε, για το blending και δεν το άκουσα και ευχαριστώ κύριε Κράμερ που μου δίνετε το λόγο πολύ σύντομα. Βεβαίως και οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν ε, μια δυνατότητα ε, χρήσης διαφόρων ταμείων, ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ένα δισεκατομμύριο λοιπόν ήδη από την ε, πρωτοβουλία συνδέοντας την Ευρώπη τη διευκόλυνση για καινοτόμα ε, νέα μέσα χρηματοδότησης, αλλά στην ερεσιμότητα θα συνδυαστεί και με το ΕΦΣΙ και άλλα τραπεζικά προϊόντα. Ε, αυτό σημαίνει ένα άνοιγμα προς τα σημεία που αναφέρατε και εσείς και σας ενδιαφέρουν. Δηλαδή, κοιτάμε περισσότερο προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, και να έχουμε και γεωγραφική ισορροπία που το πρώτο έτος λειτουργίας του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων αυτό εχόλαινε, έχετε δίκιο, και στα κράτη-μέλη που είχαν την δυσκολία να ενταχθούν. Αυτή η δυνατότητα συνδυασμού κονδυλίων, αυτό το blending, ένα χαρμάνι από διάφορα ε, ταμεία, ε, θα βοηθήσει να δημιουργηθεί ένα χαρτοφυλάκιο έργων που δεν είναι έτσι προφανή από την κλασική τραπεζική ε, δανειοδότηση να χρηματοδοτούνται. Είναι θετικά λοιπόν αυτά ως εξελίξεις και ελπίζουμε να μπορούμε ε, να υποστηρίζουμε και μάλλον να προσβλέπουμε και στη δική σας υποστήριξη στην προσπάθεια που κάνουμε στην εργασία μας με την τράπεζα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. πρόεδρε, τώρα που έχουμε λίγο χρόνο, Μήπως να κάνουμε και άλλη μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το σημείο για το blending, ε, το συνδυασμό διαφορών ταμείων είναι πολύ καλό και χαιρόμαστε που τα ακούμε όλα αυτά τα ευχάριστα. Αλλά μήπως θα μπορούσαν να μας πούν τίποτα για το SEF και use it or lose it, δηλαδή την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη και τα χρησιμοποιείς τα κονδύλια ή τα χάνεις. Γιατί ακούω ότι δεν προχωρούν έργα, γιατί δεν υπάρχουν άδειες, γιατί δεν υπάρχουν τοπικές επενδύσεις. Μήπως ο κύριος Ρόιτερς ξέρει να μας πει τίποτα, ε, να αυτοσχεδιάσει, ε, αν δεν μπορεί, κρίμα. Αλλά θα ήθελα να την κάνω αυτή την ερώτηση. Τι γίνεται εκεί. Και δεν χρειάζεται και να τα μεταφράσει κανείς γιατί τα καταλαβαίνει αυτά τα Ολλανδικά που του το λέω. Επειδή όλοι για μια ελπίδα ζούμε, γνωστό να του δώσω το λόγο και ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ευχαριστώ. Με την άδειά σας θα εξακολουθώ να απαντώ στα αγγλικά αν δεν πειράζει τον αξιότιμο βουλευτή. Αυτό το use it or lose it είναι τα χρησιμοποιήσει, τα χάνεις. Πραγματικά αυτό εντάσσεται στον κανονισμό ε, της ευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη και αν δεν προχωρούν τα έργα, σύμφωνα με τις συμφωνίες και τις συμβάσεις για τις χορηγήσεις που έχουν γίνει για κάθε έργο, τότε ε, ε, ο εκτελεστικός οργανισμός που επομίζεται με τη διαχείριση από πλευρά Επιτροπής αρχίζει η διαδικασία είτε αναστολής, είτε ανάκτησης, είτε ακύρωσης. Υπάρχουν και οι τρεις δυνατότητες για το έργο αυτό. Ε, μέχρι τώρα έχουμε κάνει δύο ε, προσκλήσεις το 2014 με επιλογή το 15 και μία το 15 με επιλογή το 16. Αυτές ε, οι δύο προκηρύξεις και τα έργα αυτά τρέχουν τώρα ε, ένα ή δύο χρόνια. Και εκεί ε, θα ήταν πρόωρο να εφαρμόσουμε αυτή την αρχή use it or lose it. Αλλά στις τελευταίες δημοσιονομικές προοπτικές, στην διάμεση αναθεώρηση θα γίνει αυτό και φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο επίκειται το 2018 να γίνει. Και ε, εν ευθέτω χρόνο τότε λοιπόν μπορεί να ανακτηθούν κονδύλια, να ζητηθούν από εκείνα που δεν αποδίδουν και δεν προχωρούν. Όπως γνωρίζετε ε, το χαρτοφυλάκιο είναι τριπλάσιο ή τετραπλάσιο ε, από αυτά που επιλέγουμε. Υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι που υποχρεωθήκαμε να τους απορρίψουμε. Και χρήματα που δεν απορροφά ένα έργο μπορούν πολύ εύκολα να τα απορροφήσουν κάποιοι άλλοι. Αυτό δεν το θέλουμε κατά ανάγκη γιατί ε, επιλέγουμε κάποια έργα ακριβώ επειδή έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα που δεν χρηματοδοτούνται και έχουν μείνει στα κρύα του λουτρού και θα μπορούσαν να υποφεληθούν. Παρακαλώ να μην με παρανοήσετε. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το κάνουμε αυτό για να πάρουμε τα λεφτά από τον ένα να τα δώσουμε στον άλλον. Δεν το κάνουμε κάτι τέτοιο. Απλώς αυτό το λέει ο κανονισμός, ότι θα πρέπει ένα έργο να αποδίδει και να ε, προχωράει σύμφωνα με τα όσα έχουν συμφωνηθεί όταν εγκρίθηκε. Δεν είναι μαθηματικό ότι χρειαζόμαστε 10-20% να τα πάρουμε πίσω. Υπάρχει στενή παρακολούθηση όλων των έργων για να δούμε πώς αποδίδουν. Και τα χρήματα που θα επιστραφούν, θα, ε, μάλλον αυτά που αποκομίζουν θα πρέπει να επανεπενδύονται. Ευχαριστώ σχεδόν τελειώσαμε τη σημερινή ε, συνεδρία. Να σας πω μόνο την προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. 13 Οκτωβρίου, η ψηφο... 14 Οκτωβρίου, 14 ε, για τις τροπολογίες. Εδώ θα ψηφίσουμε στις 10 Νοεμβρίου, στην Επιτροπή Οικονομικών στις 29 Νοεμβρίου, ενώ στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Αυτά. Εδώ ολοκληρώνεται τη σημερινή μας συνεδρίαση. Ακολουθούν οι συντονιστές θα ήθελα να παρακαλέσω εκείνους που δεν συμμετέχουν συνεδρίαση των συντονιστών που δεν επιτρέπεται δηλαδή να αποχωρήσουν. Νομίζω από χρόνο πάμε καλά και μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα. Δεν ξέρω, Λούση, μπορείς να πάρεις τηλέφωνο τον Ισμαήλ Αρτούκ να έρθει το συντονιστή σας. Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε. Να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και μετά μέσω συντονιστές. Και αν είναι παρόν ο κύριο Ρόιτερ και στη συνεδρίαση των συντονιστών θα του δώσουμε πρώτο το λόγο. Έρχεται είπαμε.